Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον υποψήφιο Επίτροπο Οικονομίας, τον κύριο Παόλο Τζεντιλόνι, και τα μέλη της Επιτροπής Εκών Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, που είναι η αρμόδια κατουσία επιτροπή για την ακρόαση αυτή. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω τα, μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι συνδεδεμένες επιτροπές, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που είναι προσκεκλημένες επιτροπές. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για την έγκριση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τον υποψήφιο επίτροπο βάσει της γενικής επάρκειάς του, της προσήλωσής του στην ευρωπαϊκή ιδέα και της προσωπικής του ανεξαρτησίας. Επίσης, αξιολογεί τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει και τις ικανότητες επικοινωνίας. Όπως ξέρετε, είχαμε στείλει γραπτό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει απαντήσει επίσης γραπτό επίτροπος, ο υποψήφιος επίτροπος, και οι γραπτές απαντήσεις έχουν σταλεί στα μέλη μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες. Η Επιτροπή μάλιστα Νομικών Υποθέσεων δεν έχει γύρει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης. Να σας εξηγήσω τώρα συντομία την ε, οργάνωση, τα διαδικαστικά. Ο υποψήφιος επίτροπος καλείται να κάνει μια αρχική προφορική δήλωση που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στη συνέχεια και στο τέλος συνεδρίασης θα έχει 5 λεπτά για τα καταληκτικά του σχόλια. Μετά την εισαγωγή του υποψηφίου επιτρόπου θα έχουμε χρόνο για την υποβολή 25 ερωτήσεων από ευρωβουλευτέ. Θα γίνονται σε 5 λεπτά ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση του οριστέντα επιτρόπου και σε περίπτωση που υπάρχει επερώτηση δεν θα πρέπει αυτή να υπερβαίνει το ένα λεπτό και μονόλεπτη θα είναι και η απάντηση του υποψήφιου επιτρόπου. Ο πρώτος γύρος θα παρτίζεται από επτά ερωτήσεις και θα υποβληθούν από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο δεύτερος γύρος από 18 ερωτήσεις ακολουθεί τη γενική κατανομή ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων συμπεριλαμβανομένου και ενό εκπροσώπου μη εγγεγραμμένων μελών. Η διερμηνία προβλέπεται σε 23 γλώσσε, οπότε όλοι οι ομιλητέ μπορούν να χρησιμοποιούν τη μητρική του γλώσσα. Απλώ να σα υπενθυμίσω ότι επειδή οι ομιλίε του μεταφράζονται, μην μιλάτε πολύ γρήγορα για να σα προλαβαίνουν και οι διερμηνείς. Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίση είναι δυνατόν ε, να λάβετε μαγνητοσκοπημένη ε, μαγνητοσκοπημένο βίντεο της ακρόασης στην ιστοσελίδα επίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο τον κύριο Τζεντιλόνι για μια προφορική δήλωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Presidente, signore deputate, signori deputati, sono davvero onorato di essere qui con voi stamattina. In quasi vent'anni di esperienza parlamentare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 όταν ε, συμβεί αυτό, ε, ε, όταν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ελπίζω να επιβεβαιωθώ ως Επίτροπος. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω μια διαδικασία ανάκαμψης. Οι δύο είναι οι όροι, φιλοδοξία και συνεργασία και συνένεση. Θέλουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα στο οποίο να συμφωνούμε όλοι και να ξαναρχίσουμε την προσπάθεια. Δεν έχουμε ξεπεράσει τι δυσκολίε τη οικονομική κρίση και είχαμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη τι έχουμε μπροστά μα. Το Brexit με τους αστάθμιτους παράγοντες που δεν έχουν καθορίσει ακόμα το αποτέλεσμα, ότι ε, υπάρχει ε, ε, εντύπωση και η έλλειψη εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο μέρο των συμπολιτών μα απέναντι στην Ένωση. Υπάρχουν γεωπολιτικέ αβεβαιότητε και ανασφάλεια και ε, βεβαίως οι τεχνολογικές εξελίξεις που φέρνουν νέες δυνατότητες και δημιουργούν φόβους και σύγχυση ως προς την ταυτότητα. Φυσικά οι προκλήσεις αυτές ε, αντιμετωπίζονται από τις διάφορες χώρες σε διαφορετικό βαθμό. Ωστόσο υπάρχει διαφορά μεταξύ οικονομικής κρίσης σαφώς και της ε, ανεπαρκούς κοινωνικής και περιβαλλοντικής της βιωσιμότητας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δηλαδή θέλουν απαντήσεις. σκεφτούμε τα παιδιά που έχουν γεννηθεί αυτή τη χιλιετία. Ξέρω ότι δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε ε, τους, ε, τις προσδοκίες τους για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Θέλουμε όλοι να βεβαιωθούμε ότι για πρώτη φορά στην Ένωσή μας υπάρχει μια, να μην υπάρχει μια γενιά που έχει λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχαν οι γονείς τους, μητέρες και πατέρες. Η δική μου γενιά ε, πήρε πολλά από την Ενωμένη Ευρώπη και εγώ είχα την τιμή να το θυμίσω. Στην πόλη μου, τη Ρώμη, με την επίσημη δήλωση όπου η κρατών κρατών και κυβερνήσεων και ο, οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων γιόρτασαν τα 60 χρόνια από την υπογραφή των συνθήκων. Η ειρήνη, η ελευθερία και απελευθέρωση από τι δικτατορίε, τα ατομικά δικαιώματα, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το τέλο του διχασμού τη Ευρώπη, που από σήμερα στι 3 Οκτωβρίου περνάει σε μια σημαντική φάση και θυμίζουμε σήμερα κατά την επέτειο τη επανένωση τη Γερμανία. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πετύχαμε μα δείχνουν ότι πρέπει να να είμαστε φιλόδοξοι στο πρόγραμμά μας για να πετύχουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να πάυσουμε όταν ε, την κίνησή μας, όταν γύρω μας τα πάντα κινούνται. Αυτά ήταν τα λόγια ενό από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ζαν Μονέ. Και είναι επίκαιρα περισσότερα από ποτέ σήμερα. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη και είμαι βέβαιος ότι σε αυτόν τον ορίζοντα φιλοδοξιών ε, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν να είναι πραγματικά οι πιο ε, ε, εργατικοί και άοκνοι Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη με ταπεινοφροσύνη και τόλμη. Η δέσμευσή μας για την Ευρώπη ήταν πάντοτε στο κέντρο του πολιτικού μου έργου και προσανατολίζει τη δουλειά μου στην Ιταλική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Είναι ε, ιδιαίτερος ενθουσιασμός μου για την πρόκληση αυτή, επειδή είμαι και Ιταλός και αισθάνομαι και Ευρωπαϊκός. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Στι πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη, η πρόεδρο, η οριστήσα πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι η Ευρώπη θέλει να περάσει σε μια μετάβαση για έναν υγιή πλανήτη και ένα ψηφιακό κόσμο. Η Ευρώπη μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής μόνο αν φέρει του καλύτερου ε, να συνεργαστούν και δημιουργήσει μια κοινωνική ε, οικονομία και ένα μοντέλο. Αυτό είναι η γραμμή και η αρχή που θα με οδηγήσει. Θέλω να εργαστώ στο πλαίσιο τη Επιτροπή. Επιτροπής με τον κύριο Ντομπρόφσκη και τα άλλα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων για να αντιμετωπίσω τις θεμητές προσδοκίες των Ευρωπαίων, την ευημερία, τη σταθερότητα και την προστασία. Ο, ο δικός μου χάρτης ως Επιτρόπου για την οικονομία θα βασιστεί στις ε, προτεραιότητες που έχει ε, καθορίσει στην επιστολή της, ε, στην επιστολή Ερμοδοτήτων και η Πρόεδρος Φόντερ Λάιον. Ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργείται εδώ και 25 χρόνια. Εδώ ε, όλοι αισθανόμαστε μια κατεπίγουσα ανάγκη για να εργαστούμε και να προστατεύσουμε το κλίμα μας. Θα χρειαστούν πρωτοβουλίες σε πολλά μέτωπα. Την βιώσιμη και συμμετοχική ε, ανάπτυξη. Εδώ θέλουμε να έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τα κράτη-μέλη για ε, συστηματικό και εντατικό διάλογο με τις κυβερνήσεις, του κοινωνικούς εταίρου και του πολίτε. Ω μέλο ε, της, ως μέρος της διαδικασίας οικονομικής εποπτείας θα κοιτάξουμε να ενσωματώσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό εξάμεινο χωρίς να χάσουμε την την κεντρική σημασία και την ανάγκη για αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε. Όμω, ε, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει και κοινωνική βιωσιμότητα. Οι ανισότητε εντείνονται και επηρεάζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μα μοντέλο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν με πυγμή και κατεπηγόντω. Θα πρέπει να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των φύλων, τη ανισότητε των φύλων και αυτό θα είναι βασική προτεραιότητα. Μια βασική δράση θα είναι επίση το σύστημα αντασφάλισης για τους ανέργους, το σχετικό πρόγραμμα. Ε, και εδώ ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που το ζητούσατε εδώ και καιρό. Πολιτικός δεν θα είναι απλό να το πετύχουμε. Όμως μαζί μπορούμε να πετύχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να προσφέρει προστασία στους πολίτες ε, τη στιγμή που περνάνε δύσκολες στιγμές στη ζωή τους θα φροντίσω να παρακολουθώ την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν ε, εύρυθμα, εύρυθμη διαχείριση των ε, δημοσιονομικών και θα υπάρχουν και ε, αποφάσεις ευελεξίας κατά περίπτωση όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την δημοσι... να αλλάξουμε τη δημοσιονομική μας τάση για να καθοριστεί σωστά η γραμμή της ανάπτυξης και να τονώσουμε τις επενδύσεις. Στην εφαρμογή των κανόνων μας θα επικεντρωθώ και στη μείωση του δημοσίου χρέους ως κάποιος που πραγματικά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επίδραση που μπορεί να έχει το δημόσιο χρέος σε δύσκολες στιγμές και να φέρει αποσταθεροποίηση. Εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ε, Επαρκέ φορολογικό ε, πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε και την επιβράδυνση που μπορεί να γνωρίζει η οικονομία μα βεβαίω, το Σύμφωνο ε, ανάπτυξη και σταθερότητα δεν είναι τέλειο. Θα εκμεταλλευτώ λοιπόν την ευκαιρία που θα μα δώσει αναθεώρηση του ξάπτυχου και του δίπτυχου για να σκεφτούμε ποιο είναι ο κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε βασιζόμενο στα διδάγματα του παρελθόντο και λαμβάνοντα υπόψη τι συνεισφορέ του Ευρωπαϊκού Σχετικού Συμβουλίου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Θα ξεκινήσει επίσης το δεύτερο μέρος του Invest EU και ε, το βιώσιμο πρόγραμμα για τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Η μετατροπή της οικονομίας μας απαιτεί επενδύσεις. Επενδύσεις για να πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση, για να γίνει πιο πράσινη η οικονομία μας και να πετύχουμε τους στόχους μας για την απελαγή από τον άνθρακα. Οι επενδύσεις για την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση είναι σημαντικέ. Οι επενδύσεις για τις βιώσιμες υποδομέ για τι για τις ε, κοινωνικέ και κοινωνικέ επενδύσεις μάλλον. Χρειάζεται δράση η οποία να ενισχύσει το ενιαίο μα νόμισμα, το κοινό μα νόμισμα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την νομισματική και οικονομική ένωση. Μία προτεραιότητα για την σα πρόεδρο και για μένα τον ίδιο. Θέλω λοιπόν να αποτίσω φορό τιμή στο σώμα σα και στην Επιτροπή σα όλο ιδιαίτερω για του φιλόδοξου στόχου σα σε αυτό τον χώρο. Πραγματικά χρειάζεται μία μεγάλη ε, αλλαγή στην σταθερότητα, για να υπάρχει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην Ευρωζώνη, να ενισχύσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ευρώ ε, διεθνώ, που είναι γεωπολιτική προτεραιότητα για όλου μα. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, 74% των πολιτών συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να καταπολεμήσει τη φοροαπάτη. Είμαι αποφασισμένος να εργαστώ προς ένα δίκαιο σύστημα φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να βεβαιωθώ ότι η φορολογία πραγματικά συμβάλλει στην, ε, στο Green Deal, αυτή την ε, πράσινη ε, νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν ένα φορολογικό πλαίσιο για την Ευρώπη ώστε να καθοδηγήσουμε την ε, συμπεριφορά των παραγωγών, καταναλωτών και χρηστών για μια οικονομία ουδέτερη ως προς τις κλιματικές αλλαγές. Θα προβλέψω μια σειρά από μέτρα που να συμπεριλαμβάνουν και την οδηγία για τους ενεργειακούς φόρους ώστε αυτά να ευθυγραμμιστούν με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και θα κοιτάξουμε να εργαστούμε σε έναν φόρο για τον άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα σύνορα ε, βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι κοινωνικός και οικονομικός ισόρροπο και θέλουμε να αποτιμήσουμε και την ε, ε, ε, αξία των ρητρών για την μετάβαση και βάσει στις συνθήκες, ώστε να υπάρχει και δυνατότητα ε, της έγκρισης αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία στη διαδικασία της συνομοθεσίας. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα του διεθνούς εταιρικού φόρου, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Όλοι κατανοούν ότι το σύγχρονο σύστημα είναι πλέον ξεπερασμένο. Η μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόσταση ε, του μεταξύ ε, πού παράγεται η οικονομική, το οικονομικό κέρδος, το όφελος και πού καταβάλλεται ο, φόρος. ο φόρος. Αυτό διαστρεβλώνει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών και τελικά δεν επιτρέπει να ε, λύσουμε το απαραίτητο φοροσπρακτικό εισόδημα. Εδώ λοιπόν ε, κοιτάζουμε στο G20, στηριζόμενοι από τον ΩΣΑ, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να σταθμίσουμε πώ έχουν προχωρήσει τα πράγματα διεθνώ. Αν δεν υπάρξει καμία συμφωνία διεθνώ, πραγματικά θέλω να οδηγήσω όλε τι προσπάθειε προ έναν δίκαιο ευρωπαϊκό φόρο και μια κοινή εταιρική φορολογική βάση. Τρίτη μου προτεραιότητα είναι να συνεχίσω να πολεμώ κατά τη φοροαποφυγή και φοροαπάτη. Κάτι που ε, πραγματικά διαστρεβλώνει και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στο φορολογικό σύστημα. Οι φορολογούμενοι θέλουν να πληρώνουν βάσει των νόμων και να υπάρχει και τιμωρητική ε, αντίδραση σε όσου δεν πληρώνουν, δεν καταβάλουν το φόρο τους. Τέλος, θα είμαι περήφανο να αναλάβω κατά της Τελωνιακή ένωσης Ένα βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ένα στοιχείο που διαφυλάσσει την ενιαία μας αγορά. Πολλοί θεωρούν την Τελωνιακή Ένωση ω κάτι δεδομένο. Ωστόσο, υπάρχουν εντάσεις σε όλο τον πλανήτη σε σχέση με τα θέματα του εμπορίου, την ασφάλεια και την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου το ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτό απαιτεί μια ισχυρότερη τελωνιακή ένωση. Θέλω λοιπόν η τελωνιακή ένωση να έρθει στο προσκήνιο και να περάσει στο επόμενο επίπεδο αποτελεσματικότητα. Δεν είναι μόνο όμω τα σχέδιά μου, αλλά και όλε οι προτεραιότητε που αναφέρονται από τον οριστήσα πρόεδρο ε, στην επιστολή που θα αποτελέσουν μια σαφή βάση για να ε, αλλάξουμε και το βαθμό αξιοπιστία των στατιστικών μα δεδομένων. Θέλουμε να είναι ανεξάρτητη Eurostat και να μπορεί να σταθεί δίπλα στι ε, διεθνεί ανεξάρτητε αρχέ. Θέλουμε η Eurostat να παραμείνει ένα, αξιο, ένα αξιόπιστο σημείο αναφορά για τα στατιστικά μα δεδομένα και τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε για ε, την ε, οικονομία και την Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ θύμισα ορισμένα μόνον σημεία, τους πρωταρχικούς στόχους που εφόσον εγκρίνεται την, ε, ε, τον διορισμό μου θα χαρώ να επιδιώξω στη θητεία μου. Σε πολλές περιπτώσεις για να τα πετύχω έχω ανάγκη από τεράστια πολιτική δράση και αγώνα. Θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες για να ε, προκρίνουμε τελικά τι ε, κοινέ συμπεφωνημένε λύσει. Θέλω να δω τι διαφορετικέ απόψει μεταξύ διαφορετικών πολιτικών οικογενειών, χωρών, διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη. Όμω θέλω όλοι μαζί να αποφύγουμε οι διαφωνίε μα, να δημιουργήσουν περισσότερε προκαταλήψει και τελικά να γίνουν τροχοπέδι στο να επιδιώξουμε την ε, ε, γοργή πορεία μα προ την αλλαγή που χρειάζεται. Θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Η πολιτική μου εμπειρία δεν είναι σύντομη. Ε, και είναι σαφές ότι πρόκειται για την ανάγκη να εξεύρουμε λύσεις, να διαπραγματευτούμε συμβιβασμούς και να εργαστεί η Επιτροπή ως κολέγιο, σε μορφή σώματος συλλογικού. Θα πρέπει να επιδιώξουμε και το πολυτιμότερο όμως αγαθό, ε, την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και ενδιαφερομένων. Εσείς θα είστε για μένα ένα σταθερό σημείο αναφοράς, με ε, τακτικές και συστηματικές διαδικασίες διαλόγου. Θα φροντίζω να ενημερώνω την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ προτού ληφθεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα εργαστώ μαζί σας όλος ιδιαιτέρως για τις νέες νέες που έχει ε, καταδείξει και η πρόεδρο Φόντερ Λάιεν. Είναι κεντρικό ε, ο χαρακτήρα ε, τη σημασίας του ρόλου συνεργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε να σεβαστούμε όλους τους θεσμικούς κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολιτική επιλογή σε καιρού όπου σε διεθνέ επίπεδο η προάσπιση της δημοκρατίας, της φιλελεύθερη και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έχει γίνει πλέον ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο. Σα ευχαριστώ πολύ και περιμένω τι ερωτήσει σα. Σας ευχαριστούμε κύριε Τζεντιλόνη. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ξεκινούμε από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Πρώτος ε, ο Μάρκος Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνη πολλά τηλεφωνήματα έλαβα από τη Ρώμη πόσο εξαιρετικό υποψήφιο είσαστε. Μόνο ο Πάπα δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Ωστόσο, θα ρωτήσω κάτι. Το κρίσιμο ερώτημα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πώς το βλέπεις. Ε, στην προηγούμενη Ιταλική κυβέρνηση είπατε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, αλλά το πώς αντιλαμβάνονται οι αγορές, ε, το ότι αγνοούμε τους κανόνες. Ε, θα συμφωνήσω με αυτό. Ωστόσο, έχετε ε, επικρίνει επίσης το σύμφωνο. Η νέα κυβέρνηση της χώρας σας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας σας, αναφέρεται κυρίως στην έλλειψη ευελιξίας του συμφώνου και προβλέπεται όχι μόνο αν ονομαστική αύξηση του ελλείμματος, αλλά και ουσιαστική αύξηση. Ε, κάτι στο οποίο δεν είμαστε πια, για το οποίο δεν είμαστε πια προετοιμασμένοι. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς το σύμφωνο και πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή τήρηση των κανόνων και στο, στον Ιταλικό προϋπολογισμό. Uh, well, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φέρμπερ. Ευχαριστώ και όσους σας πήραν τηλέφωνο από τη Ρώμη. Νομίζω ε, ότι είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Έχουμε τους κανόνες μας, έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πρέπει να το εφαρμόσουμε. εντός του συμφώνου υπάρχει ευελιξία και αυτό δεν είναι παραχώρηση προς τη μία ή την άλλη χώρα. Είναι κάτι που περιέχει το σύμφωνο από μόνο του. Δεν θα σχολιάσω το Ιταλικό σχέδιο προϋπολογισμού, διότι παρεμπιπτόντως δεν το έχουμε ακόμη. Προσχέδιο προϋπολογισμού θα έχουμε σε 12 μέρες από σήμερα. Και θα το εξετάσω με την ίδια προσοχή, με την ίδια διάθεση για διάλογο και την ίδια σοβαρότητα ε, σε σχέση με τους κανόνες ε, που ε, θα δώσω και στα άλλα 26 κράτη-μέλη. Κύριε Φέρμπερ, Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής αν είναι δυνατόν. Δεν θα εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Εγώ θα είμαι επίτροπος οικονομικών υποθέσεων. Και με την ιδιότητά μου αυτή θα ασχοληθώ με όλα τα προσχέδια προπολογισμού όταν αναλάβω τα καθήκοντά μου, εφόσον επιβεβαιώσετε εσείς, ε, ε, ε, εφόσον εγκρίνετε την υποψηφιότητά μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζεντιλόνι. Υπάρχει το πρωτόκολλο, το πρόσθετο πρωτόκολλο στο σύμφωνο, που πιάνει μόλις δύο σελίδες. Το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ερμηνεία των κανόνων είναι πάνω από 100 σελίδες. δεν ε, θα σας ρωτήσω τώρα αν ανάμεσα στο βήμα 1 και το βήμα 17 θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το βήμα 9, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε απλούστευση ώστε τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν καλύτερα τους κανόνες και όχι το κάθε κράτος μέλος ε, να επιλέγει κανόνες ε, όπως το βολεύει. Δεν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια στο σύμφωνο για να είναι και πιο ε, εύκολη και σαφής η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ε, μη τήρησης των κανόνων. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι καθόλου απλοί του SGT, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εκτιμώ πολύ την συνεισφορά που δόθηκε που ε, ε, ήταν συγκεντρωμένη σε τρία ε, σημεία που ήταν εύκολο να εφαρμοστούν και ήταν αντικυκλικά. Τώρα, όπως γνωρίζετε, αναθεωρούμε τώρα την δέσμη των 2 και 6 νομοθετικών μέτρων αντίστοιχα, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ε, θα είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Θα έχουμε νομοθετικές αλλαγές ή θα ερμηνεύσουμε με πιο απλό τρόπο τους κανόνες μας. Αυτή θα είναι μια σημαντική συζήτηση στην οποία θα συνεισφέρω. Σας ευχαριστούμε. Ο Χώνας τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε υποψήφιο επίτροπε. Φαίνεται ότι η Ευρώπη έχει μια επιβράδυση της οικονομίας της. Μια επιβράδυση όταν ταυτόχρονα η νομισματική πολιτική φαίνεται ότι έχει τα όρια της. Και είναι προφανές όπως είπατε και εσείς ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Γι' αυτό όμως ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε προηγουμένως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί ο στόχος και το όραμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών. Και καλά κάνει βέβαια. Αλλά η ίδια προσπάθεια ε, που αφιερώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη για τη μείωση των ε, ελλημάτων των δημοσιονομικών θα πρέπει ε, να, την, να κάνει αντίστοιχε προσπάθειες για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Ε, όπως είπατε, έχει αντικυκλικό χαρακτήρα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό όμως προϋποθέτει την ε, ισχύ της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να βοηθήσει τα κρατημέλη να βελτιώσουν τον κύκλο τους. Πώς προτίθεστε να αναθεωρήσετε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ναι, όντως παρατηρούμε μία επιβράδυνση της οικονομίας μας, όπως είπατε κύριε Φερνάντες, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όντως, παρατηρούμε μία επιβράδυση της οικονομίας. θα έχουμε τις οικονομικές μας προβλέψεις περίπου σε ένα μήνα, σε αρχές του Νοεμβρίου. Και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να αντιληφθούμε τις διαστάσεις αυτής της οικονομικής επιβράδυσης και τη διάρκεια που θα έχει για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε περί δημοσιονομικού προσανατολισμού. Πάντως, γενικώ, συμφωνώ μαζί σας ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στη μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων, αλλά να μεριμνά και για την ανάπτυξη. Και μάλιστα επιδιώκει μια συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. Γιατί αν έχουμε μόνο τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής, δεν αρκεί αυτό. Δεν μας αρκούν μόνο τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής. Γενικώ δεν αρκούν, αλλά ειδικώ στους καιρούς αυτούς που αντιμετωπίζουμε μια οικονομική επιβράδυση, θα πρέπει να προσθέσουμε στη νομισματική πολιτική μια πιο συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική. Με τις διαφοροποίησεις, τις προφανείς διαφοροποίησεις μεταξύ των κρατών μελών και ταυτόχρονα θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαιτέρως στις επενδύσεις. Νομίζω ότι έχουμε πολλά μέσα και εργαλεία στο πρόγραμμα της Ursula von der Leyen για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και τις προσπάθειές μας να προσελκύσουμε επενδύσεις και ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους και οδησηγητές για την απόφασή τους που κατέσαν δυνατή την έγκριση του προγράμματος Invest EU, που θα είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό την επόμενη πενταετία. Επερώτησε ο κύριος Χώνας Φερνάνδες. Μάλιστα κύριε υποψήφια, το θέμα είναι ότι εκτός της αναγκαίας αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να υλοποιήσουμε μια σφαιρική πολιτική ε, πιο αντικυκλική στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειαζόμαστε και κάποια μέσα για την Ευρωζώνη, κάποια κεντρικά ε, μέτρα και μηχανισμούς για την Ευρωζώνη που θα συμπληρώσουν τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές ώστε να δώσουν μια επιπλέον ε, δημοσιονομική θέση στην Ευρωζώνη. Και οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και η δέσμευση τη ε, κυρία Φόντερ Λέιν για την αντασφάλιση για, την, για τι παροχέ ανεργία ή η πιθανοτητα προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Γίνονται παράλληλα αυτέ οι συζητήσει. Πώ ε, βλέπετε την ιδέα ενό κεντρικού οργάνου, ώστε οι εθνικέ πολιτικέ που αναθεωρούνται στα πλαίσια σταθερότητα και ανάπτυξη να έχουν ένα, ένα πιο γενικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα με προτάσεις για τη βελτίωση του κύκλου, του οικονομικού του κύκλου. Τζεντιλόνι. Έχουμε ακούσει πολλές ε, προτάσεις τον τελευταίο καιρό και έγκριτες προσωπικότητες να προτείνουν ότι χρειάζονται και κάποια σταθεροποιητικά εργαλεία στην νομισματική μας ένωση. Αυτό ε, είπε και πριν από λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος της ΕΚΤ, ο Δράγκη. Πολύ συχνά αναφέρεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τον ΩΣΑ. Αλλά είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν πολιτικές ε, διαφορές και διαφωνίες μεταξύ των κρατών μέλων. Η σαν πρόεδρος επισήμανε κάποια χρήσιμα εργαλεία κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης των Παροχών Ανεργίας. Το δεύτερο είναι το Δημοσιονομικό Μέσο Σύγκλησης και Ανταγωνιστικότητας. Έχουμε όμως και άλλες προτάσεις περσινές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι δεν είναι θα πρέπει να τις ε, απορρίψουμε. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά έχοντας υπόψη ότι το μέλλον της ΟΝΕ έγκυται στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και με κάποια εργαλεία σταθεροποίησης. Σας ευχαριστώ. Ο Λουίς Καρικάνο από το Renew Europe. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλόνε. Τζετιλόνη. Θα ήθελα να ε, συνεχίσω αυτό το θέμα των εργαλείων σταθεροποίησης και την ε, αντασφάλιση παροχών ανεργίας που πρότεινε η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις. Νομίζω ότι είναι μια μορφή πολιτικής σταθεροποίησης αυτή η πρόταση. Ε, μια ασφάλεια για την ανεργία είναι ένα αντικυκλικό μέτρο που μπορεί να βοηθήσει τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Αλλά βέβαια ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λέμε. Αυτά θα πρέπει να προσέξουμε. Ποιες είναι λοιπόν οι δικές σας ιδέες και απόψεις για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτό το σύστημα αντασφάλισης παραχών ανεργίας, ώστε να αποτρέψουμε κάποιους κινδύνους που προβληματίζουν πολλούς και εμάς στο Renew Europe, ώστε να μην έχουμε μόνιμες μεταβιβάσεις, να μην έχουμε ηθικό κίνδυνο και να ενταχθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Παραχών Ανεργία στα εθνικά συστήματα επιδομάτων ανεργίας. Ποιες είναι οι ιδέες σας ε, για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα αντασφάλισης παραχών ανεργία, ώστε να αποτρέψει τους κινδύνους που προανέφερα. Σας ευχαριστώ κύριε Γαρικάνο. Η πρόταση αυτή έχει ένα διτό σκοπό. Και φυσικά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τον πρωταρχικό σκοπό αυτής της πρότασης, που είναι ο κοινωνικός σκοπός ενός συστήματος που ενισχύει τα εθνικά συστήματα και προστατεύει τους ανέργους. Οπότε μέλημά μας είναι οι πολίτες. Και η πρόταση αυτή έχει ένα σαφές κοινωνικό μήνυμα και κοινωνική πρόθεση, αλλά έχει ταυτόχρονα και μία σταθεροποιητική επίπτωση. Δεν είναι μόνο εργαλείο σταθεροποίηση, δηλαδή αυτό το σύστημα αντασφάλιση παροχών ενεργεία που προτείνει η κυρία Φοντερ Λάιεν. Έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Τώρα, είπατε τι δεν θα πρέπει να είναι αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα αντασφάλιση παραχών ενεργεια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εργαλείο μόνιμων μεταβιβάσεων από χώρα σε χώρα. Επίση, αυτό το σύστημα δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει τι εθνικέ διαδικασίε διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό το μέτρο θα πρέπει να επικεντρώνεται σε εξωτερικούς κραδασμούς και να έχει μηχανισμούς ταχείας πληρωμής, ταχείας εκταμίευσης. Εγώ έχω αναλάβει τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του μηχανισμού και αυτό θα είναι το βασικό θέμα και από πολιτική και από τεχνική άποψη. Θα δούμε αν το ευρωπαϊκό αυτό σύστημα αντασφάλισης παροχών ενεργείας θα επικεντρώνεται σε δάνεια ή σε άμεση υποστήριξη των εθνικών προϋπολογισμών. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική και δεν σημαίνει ότι αυτά τα δύο σενάρια είναι αντιφατικά μεταξύ τους τελείως ή αντιμαχόμενα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο σενάριο και να το διαμορφώσουμε στη συνέχεια. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, πάντως πολύ σύντομα και φυσικά αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Επερώτηση από τον κύριο Καρικάνο. Ναι, προσβλέπουμε και εμείς σε στενή συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. ποιο είναι όμως το όραμά σας ε, για το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΟΝ. Πότε προβλέπετε να υποβάλλετε την πρόταση. Θα είναι κορυφαία σας προτεραιότητα, θα το αφήσετε για λίγο αργότερα. Πότε προτείνετε να υποβάλλετε τις μεταρρυθμιστικές αυτές προτάσεις και στην ΕΚΟΝ. Φυσικά θα ασχοληθώ αμέσως με το θέμα αυτό. Αμέσως. Τώρα το αμέσως θα εξαρτηθεί και από τις πολιτικές εξελίξεις. Αμέσως, αν μου δώσετε φυσικά την έγκρισή σας, θα εγκύψω στο θέμα αυτό με τον συνάδελφο Σμιτ και με το Συλλογικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι σαφές ότι αυτό το σύστημα Ε, με βάση ρευστότητα και δάνεια θα είναι εύκολο. Ευκολότερο τουλάχιστον, γιατί εύκολο δεν είναι τίποτα. Ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε δάνεια και ρευστότητα θα είναι πιο ταχύ στην αντίδρασή του και θα στηρι... και το θέμα της, ε, βέβαια το άλλο ζήτημα της δημοσιονομικής στήριξης είναι πιο περίπλοκο και θα έχει συνέπειες και στον στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Πάντως είπα στην αρχική μου δηλώση ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι και σε αυτό το θέμα του συστήματος αντασφάλισης παροχών ανεργίας. Ευχαριστώ. Ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους. Κύριε Τζεντιλόνι, είχαμε τα LuxLeaks και άλλα φορολογικά σκάνδαλα που έχουν βλάψει την δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά η τελευταία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνέβαλε στην επανόρθωση της κατάστασης ε, μετά από πίεση του Κοινοβουλίου. Αλλά παραμένει η άδικα χαμηλή φορολογία για κάποιους. Σκοπεύεται να υποβάλλεται σχέδιο για δίκαιη και πράσινη φορολογία που να συμπεριλαμβάνει τα εξή. Ε, μια νέα δέσμη μέτρων για αποτελεσματική φορολόγηση εταιριών, ώστε να υπάρχει ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη. Και δεύτερον, ε, μετάβαση σε ε, ενεργειακή και περιβαλλοντική φορολογία, συμπεριλαμβανομένη φορολογία επί τη κυροζήνη για τι αερομεταφορέ. Επίσης να, υπάρχει, να εφαρμόζεται η αρχή ότι ο Ριπένον πληρώνει με ε, φορολογία του διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι το θέμα της φορολογίας που επί δεκαετίες δεν θεωρεί το ιδιαίτερα σημαντικό στις πρωτοβουλίες ε, των ε, ευρωπαϊκών θεσμών για λόγους που πολύ καλά γνωρίζετε. Γίνεται όλο και πιο επίκαιρο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Εγώ λοιπόν πρέπει να εκτιμήσω αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ εύστοχα αυτά που έγιναν. Δικό μου έργο λοιπόν θα είναι να ε, συνεχίσω και να ενισχύσω τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στο θέμα αυτό. Η πρόταση που κάνατε για δέσμευση πάνω σε νέο σχέδιο δράσης θα μπορούσε να αποτελεί κατά τη γνώμη μου τρόπος για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να στείλουμε αμέσως το μήνυμα ότι ναι, είμαστε προσιλωμένοι στα θέματα αυτά. Το περιβάλλον, την, ε, τις επιχειρήσεις, ε, την ψηφιοποίηση, τη φορολογική απάτη. Θα ήταν χρήσιμο να προτείνουμε στο Σώμα των Επιτρόπων ένα σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον ε, των πολιτών μας ε, και που να λαμβάνει υπόψη και την κοινή γνώμη πάνω στο θέμα αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι ε, αυτή είναι μία προσωπική πολιτική δέσμευση. Εργαζόμαστε εντός του σώματος και ε, δουλεύουμε μέσα σε ένα διαθεσμικό πλαίσιο όπου οι αποφάσεις για την φορολογία λαμβάνονται ομόφωνα μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτή λοιπόν θα είναι μια από τις βασικές πολιτικές μας προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για την προσωπική σας δέσμευση. Πέρα από αυτό, κάποιες από τις προτάσεις της τελευταίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν μπλοκαρισμένες στο Συμβούλιο. Στις γραπτές σας απαντήσεις ε, είπατε ότι είστε διατεθειμένος σε κάποιες από αυτές ε, τις προτάσεις ε, να μην απαιτούν πια ομοφωνία, αλλά να απαιτούν πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 116 της συνθήκης. Μπορείτε να μας πείτε ήδη τώρα Ποιες από τις προτάσεις αυτές ε, σκοπεύετε να τις κάνετε αντικείμενο ε, ε, υπερψήφισης με πλειοψηφία αντί για ομοφωνία και πότε σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολύπλοκα νομικά θέματα εδώ. Εάν παραπέμψουμε στο άρθρο 116, τότε ε, παραπέμπουμε σε παρεκκλήσεις ε, όσον αφορά τις συνθήκες στην εσωτερική αγορά. Εάν λοιπόν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 116, τότε η επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να ε, συνδέονται ε, αποκλειστικά με το θέμα αυτό. Δηλαδή, θέματα περιβαλλοντικά ή φορολογίας εταιριών δεν μπορούν να, να ε, χρησιμοποιηθούν στο... δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 116. Πρέπει να υπάρχει σημαντική παρέκκληση και ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου, αλλά όσον αφορά την ε, ρήτρα ε, Πασαρέλ θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι πιο νομικά δεσμευτική από το άρθρο 116, χρειαζόμαστε όμως ομοφωνία. Ευχαριστώ. ID. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρινάλντι από την ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επιτροπή, θα μιλήσω Ιταλικά. Κύριε Τζεντιλόνι, δεν θεωρείται ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον υπολογισμό του output gap, του καινού ε, προϊόντος ε, για το σύστημα, όταν παίρνουμε τα χαμηλότερα δεδομένα για το χαμηλότερο καθαριστό εγχώριο εισόδημα και σε σχέση με τα δεδομένα του ΟΑΣΕ και των ε, διεθνών φορέων, ώστε να κρυθούν προς, το, τα χείρο των κρατικών υποδομών. Στις 30 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία κρίθηκε ένα προπολογισμό όπου γίνονται υποσχέσει για βελτίωση του 0,6% του διορθωτικού στοιχείου. Και το διορθωτικό σκέλος είναι 0,1%. Επιπλέον υπάρχει ένα 0,4% ε, αντιρεαλιστικών ε, προτάσεων για ανάκαμψη. Πιστεύετε ότι μπορούν να εγκριθούν αυτοί οι αριθμοί, ενώ ο ίδιο προπολογισμό δείχνει ότι δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνε περί δημόσιου χρέου, ιδίω στη σελίδα 9 του εγγράφου, και μήπω πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία παραπαραβάση όπω είχε ξεκινήσει και του χρόνου, και πέρσι, συγγνώμη. Και επιπλέον να ρωτήσω εάν πρόκειται να ασχοληθείτε με το πρόβλημα των τεράστιων εμπορικών πλεονασμάτων που έχουν σωρεύσει κάποιε χώρε, ιδίω η Γερμανία και η Ολλανδία, και που εδώ και 30 και εδώ και τρία χρόνια μάλλον, ε, διαδοχικά χρόνια, ξεπερνούν το όριο που προβλέπετε, ιδίως από το εξάπτυχο. Σας ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι. Εάν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά στα Ιταλικά λέμε το διορθωτικό σημείο μας στο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι ένα σημείο με μια κύκλωση που προβλέπεται από την Ιταλική νομοθεσία. Δεν είναι ακόμα πρόταση προπολογισμού εγκεκριμένη. Ε, οπότε επιτρέψτε μου γι' αυτό να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένω, απαντώντα σε άλλη ερώτηση. Ότι θα ασχοληθώ επισταμένος από την 1η Νοεμβρίου, εφόσον εγκριθώ για τις, με τις προτάσεις προπολογισμών και των 27 χωρών συμπεριλαμβανομένου του Ιταλικού προτάσεις που θα φτάσουν ως τα μέσα Οκτωβρίου. Και την Ιταλική πρόταση λοιπόν θα τη δούμε εντό ε, αυτής της προθεσμίας. Σε ό,τι αφορά το output gap και την ενδεχόμενη ανάπτυξη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί παρατηρητές, πολλές πολιτικές παρατάξεις οι πολιτικοί φορείς έχουν υπογραμμίσει τα τελευταία χρόνια και αυτοί οι δείκτες είναι δύσκολο να ελεγχθούν και να τους εξακριβώσει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα. Το ίδιο λέει και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η γνωμοδότηση του πρόσφατα λέει ότι θα έπρεπε να εγκρίνουμε βεβαιότερα κριτήρια, όπως έναν δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης για τις δημόσιες δαπάνες παρά κριτήρια όπως το output gap. Η, η υποθετική ανάπτυξη, η αναμενόμενη ανάπτυξη, η δυνητική ανάπτυξη, πράγμα που ακούγεται πολύ αβέβαιο. Θα το σκεφτούμε τις επόμενες εβδομάδες, τις, ε, τους επόμενους μήνες, με την ε, αφορμή της αναθεώρησης των διπτύχων και εξαπτύχων μέτρων. Χρειάζεται μια τέτοια αναθεώρηση των κριτηρίων. Ε, εξάντλησα το χρόνο μου. πάντως θέλω το δημοσιονομικό περιθώριο να υπάρχει για κάποιε χώρε και να μπορούν να το αξιοποιήσουν. Διότι οι πολιτικέ του προπολογισμού τη κάθε χώρα είναι, ε, είναι διαφορετικέ μεταξύ του, γιατί και οι χώρε διαφέρουν. Αλλά θα πρέπει το περιθώριο που θα αφήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τάχιστα. σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό, την πρόταση της 30 Σεπτεμβρίου. Ήταν στο Συμβούλιο των Υπουργών. Είναι ένα έγγραφο με, το κύριο, με τη, τη βαρύτητά του και τη σημασία του. Θα περάσει βεβαίως από τη Βουλή και θα υποβληθούν και τροπολογίες. Όμω αυτή θα είναι η βασική μορφή του. Οι τροποποιήσει θα είναι περιθωριακού χαρακτήρα. Άρα θα ήθελα να μας πείτε, εσείς όταν θα αναλάβετε ως Επίτροπος, πώς θα ερμηνεύσετε τους αριθμούς αυτούς, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση, για να το πω εντό εισαγωγικών, ε, ετύχανε διαφορετική μεταχείρισης. Και όσο αφορά το output gap, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον η μέθοδος θα πρέπει να είναι πανομοιότυπη με αυτή που χρησιμοποιεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ο ΑΣΕ. Άλλωστε θέλουμε να δούμε τι είδου σχέση θα δημορφωθεί και με τις άλλες χώρες και ιδίω με τη δυνατότητα να καταρτήσουν εκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν θα πάτε προς αυτή τη γραμμή. Ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Ρινάλντι. Για τις εκτατικές πολιτικές, πράγμα που δεν είχα χρόνο να παραπτύξω στην πρώτη μου απάντηση, να πω το εξή Βάσει των οικονομικών εκτιμήσεων και προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το καλοκαίρι, έχουμε δώσει μια ε, κατεύθυνση για μια broadly neutral fiscal stance, για μια δημοσιονομική στάση που να είναι γενικός να είναι γενικώ ε, ε, επικής, χαλαρή. Η επιβράδυνση στην ανάπτυξη, η επιβράδυνση στην ε, ανάπτυξη σκοπό έχει να δούμε αν μπορεί να ξεπεραστεί αμέσω ή να διαρκέσει. Αυτό είναι σημαντικό για να καθορίσουμε το δημοσιονομικό μας προσανατολισμό. Αυτό που θα πρέπει να δώσει ω κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι υπόλοιπες χώρες για το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Τζον Βαν από το ECR. Κύριε Τζεντιλόνι, καλή σα μέρα από εδώ. Καλημέρα σας. Ακούσαμε ήδη πολλά για το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη, δημοσιονομικού κανόνε, δημοσιονομικά ζητήματα. Είστε όμω αρμόδιος ή θα γίνετε αρμόδιος αν λάβετε την έγκριση και για την ε, Ευρωστάτ. Εκεί υπάρχει ο κανόνα ότι οι δημόσιε επενδύσει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη της, στον προπολογισμό την χρονιά τη εκτέλεση των επενδύσεων, κάτι που είναι τελείω παράλογο οικονομικά. καμία εταιρεία δεν λειτουργεί έτσι με χρονοδιαγράμματα απόσπαυση των επενδύσεων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, προωθήσουμε τις επενδύσει και να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό περιθώριο στις χώρες. Αλλάξτε λοιπόν αυτό τον κανόνα για τον υπολογισμό των επενδύσεων στον εθνικό προπολογισμό. Από τη Eurostat. Ε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. χάρη στην ερώτησή σας θα μπορέσω να κάνω και μία δήλωση που κρίνω σημαντική. Όταν ορίστηκα επίτροπος, υποψήφιος επίτροπος, και η, πρόεδρος, η εκλεγήσα πρόεδρος με ενημέρωσε ότι στις αρμοδιότητες μου θα εντάσσεται και η Eurostat, πέραν της γενικής, Γενικών Διευθύνσεων έκφυγε και ΤΑΞΟ, που ξέρετε πόσο αποτελεσματικές και ποιοτικές γενικές διευθύνσεις είναι, το μήνυμα που έλαβα και μπορώ να σας το επαναλάβω, είναι ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ένας επίτροπος, ένας επίτροπος που έχει την ευθύνη της Eurostat, την αρμοδιότητα της Eurostat, είναι να κρατήσει και να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της Eurostat. Ως προς τα κριτήρια, ως προς τους αριθμούς, ως προς τις πολιτικές. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του Επιτρόπου, να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της Eurostat. Και εγώ γνωρίζω από την εμπειρία μου στη θέση του Πρωθυπουργού και γνωρίζω ότι η πολιτική και τα μέλη της κυβέρνησης δεν είναι πάντα ικανοποιημένοι ούτε με το περιεχόμενο, ούτε με το χρονισμό των στατιστικών στοιχείων, αλλά αυτά προβλέπουν οι κανόνες. Οπότε η πρώτη μου αντίδραση στην ερώτησή σας θα ήταν ως αρμόδιος επίτροπος για τη Eurostat. Εγώ δεν θα ήθελα να επηρεάσω τα κριτήρια που αυτόνομα καθορίζονται. Θα το συζητήσει το Κοινοβούλιο, θα το συζητήσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, αλλά όχι, δεν θα το αποφασίσει ο αρμόδιος επίτροπος για τη Eurostat το αν τα κριτήρια αυτά είναι σωστά ή όχι. Επερώτηση. Και τα δημοσιονομικά θέματα έχουν σχέση με τη φορολογία. Διάβασα στις γραπτές σας απαντήσεις ότι είστε υπέρ μιας φορολογικής εναρμόνισης και αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρ και της ειδικής πλειοψηφία για φορολογικά ζητήματα. Κάτι που σημαίνει, με απλά λόγια, ότι θα είστε πιο ευνοϊκός προς τις μεγάλες χώρες και παρά στις μικρές. Τι θα κάνετε ως προς τα εύλογα ε, συμφέροντα των μικρών χωρών για τα φορολογικά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να επιδιώξω συνένεση. Και νομίζω ότι αυτό απαιτείται από έναν Ευρωπαίο Επίτροπο και ιδιαίτερα για φορολογικά ζητήματα που έχουμε, πέραν του άρθρου 116, έχουμε και τον κανόνα της ομοφωνίας για τα φορολογικά θέματα. Και γνωρίζετε την τελευταία πρόταση για σημαντική ψηφιακή παρουσία που επιβλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε, αν θυμάμαι καλά, από 24 χώρες και όχι από 27. Προς το παρόν, ε, η πρόταση αυτή έμεινε στον πάγο. Προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Οπότε, δεν έχει σημασία αν κάποια χώρα είναι μεγάλη ή μικρή σε ό,τι αφορά τον κανόνα της ομοφωνίας. Έχουμε την ε, ρήτρα ε, την παθητική, έχουμε το κοινοβούλιο, την κοινή γνώμη, το άρθρο 116. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ε, ιδέα να αποφύγουμε μία απόφαση για τη φορολογία. Η Μανώ Μομπρή έχει το λόγο, από την ΚΟΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Τζαντιλόνη. Θέλω και εγώ να μιλήσω για τα θέματα τη ε, φόρου που νομίζω ότι θα μα απασχολήσουν πάρα πολύ. Δεν θα σα απαριθμίσω τώρα τα σκάνδαλα φόρου φορολογικών παραδείσων, τα Panama Papers, τα διάφορα papers, τα Lux Leaks και ούτω καθεξή. Εδώ εμπλέκονται πολλέ πολυεθνικέ εταιρείε και μάλιστα μερικέ που τι γνωρίζετε πολύ καλά ε, λόγω του χαρτοφυλακίου αρμοδιοτήτων σα ε, πριν αναλάβετε και ω Επίτροπο την Amazon ή την LVMH όπως λέγεται, ε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφύγει το φορολογικό σύστημα και Κάποιες χώρες, ε, ε, ε, ο Παναμάς και οι Βερμούδες, είναι ένα πολύ γρήγορο, ένα πολύ γρήγορο πέρασμα μεταξύ πολλών άλλων από τον κατάλογο με τους φορολογικούς παραδείσους. Η Oxfam, που θα γνωρίζετε, σε συνεργασία με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που θα πρέπει να τις έχετε δει και εκτός κτηρίου, είχαν διαδηλώσει, το, μια δήλωση το πρωί, για να ζητήσουν να συμπληρωθεί ο κατάλογος αυτός των φορολογικών παραδείσων, που έχει πολλές ελλείψεις και που υπήρχε και στο την έκθεση της Επιτροπής ε, TAX 3 διότι είναι διαφανή και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται δεν είναι σαφή. Δεν ξέρουμε πώ τελικά κάποιε χώρε απομακρύνονται από τον κατάλογο αυτό μετά από κάποιο διάστημα. Πώ θα κοιτάξετε τον κατάλογο λοιπόν αυτό χωρί πολιτικού παρεμβατισμού, πώ θα ε, φορολογήσετε καταλήλω του μεγάλου χρηματοοικονομικού ε, ομίλου και πώ θα δείτε τι μεγάλε αποφάσει φορολογικού χαρακτήρα που μπορεί να είναι επιζήμιε, ώστε να υπάρχει και δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των ε, χωρών και εκτό συνόρων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κυρία Ομπρή, σε ό,τι αφορά το δικό μου το χαρτοφυλάκιο, και ότι εγώ χρωστούσα, έχω καταβάλει ό,τι έπρεπε και έκανα και όλες τις δηλώσεις όπως ε, ως δει, ε, προτού ε, αναλάβω Έστειλα ό,τι χρειαζόταν και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν ήμουν εκατομμυριούχο έτσι κι αλλιώ. Ε, βάσει τη Ιταλική νομοθεσία σίγουρα. Ε, Πάντω πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας και αν γίνεται και αποτελεσματικότεροι από ό,τι πριν για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων. Τώρα, αυτά που κάναμε και αποφάσει που πήραμε τα τελευταία χρόνια να μην είχαν ε, καμία αποτελεσματικότητα, λέτε. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να προασπιστώ κάτι που έκανα εγώ προσωπικό τόσο ή άλλος, διότι δεν ήμουν εγώ εδώ. Νομίζω όμως το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να είναι υπερήφανο, γιατί προ, προ, βήματα προόδου έγιναν. Και ο μαύρος κατάλογος που αναφέρατε, ο αρνητικός αυτός κατάλογος, σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί, αλλά μπορώ και εμέσως ως πρώην Υπουργό Εξωτερικών να σας το διαβεβαιώσω. Σε πολλές χώρες του κόσμου η ήπια ε, εξουσία, για να το πω έτσι, το soft power αυτό του αρνητικού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σοβαρή επίδραση. Έχει αποτέλεσμα. Αναγκάζει πολλούς να μεταβάλουν τη στάση τους, ε, αυτών που έχουν ε, ιδιαίτερα φορολογικά συστήματα. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολλά και μπορούμε να τα κάνουμε ε, μαζί, σε συνεργασία. Κυρία Τζεντιλόνη... Δεν λέω ότι υπήρχε χαρτοφυλάκιο ε, εκατομμυρίων. Βέβαια για την Amazon μιλάμε για εκατοντάδες ε, ε ευρώ, εκατομμύρια ευρώ. Όμω ελπίζω ότι αυτό δεν θα σα αποθαρρύνει από το να ασχοληθείτε με το κέρδο αυτών των επιχειρήσεων μελλοντικά. Πάντω, λέτε ότι για τον αρνητικό κατάλογο και του φορολογικού παραδείσου ε, θα υπάρξουν συνέπειε. Τι θα γίνει όμω με τα ευρωπαϊκά κράτη, όπω η Ιρλανδία και το Λεξεμβούργο. Πώ μπορεί να είναι αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δέχεται στου κόλπου τη του χειρότερου φορολογικού παραδείσου του κόσμου. Και ο συνάδελφο που πήρε το λόγο προηγουμένω να μην ξεχνάει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτοί που μπλοκάρουν τι αποφάσει δεν είναι οι μεγάλε χώρε, είναι οι μικρέ, όπω η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Όπου το βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου ε, φορολογικού ανταγωνισμού, που είναι επιζήμιο μάλιστα για τι περισσότερε χώρε. Τι θα κάνετε εσεί λοιπόν για αυτέ τι ε, επιζήμιε φορολογικέ αποφάσει, τι θα κάνετε για τι εταιρείε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, δεν πρέπει να ζητήσετε να εξετάζονται βάσει των ίδιων κριτηρίων ε, τα ευρωπαϊκά κράτη ή για θέματα μπόνους ας πούμε. Μιλάμε για θέματα που έχουν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Ε, φορολογική διαφάνεια. Θα ε, αλλάξετε το σύστημα υποβολής εκθέσεων ένα χώρα και, ώστε να είναι και δημοσίως γνωστό. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αποδεχτεί Ε, μια επιθετική πολιτική φορολογική, ε, μια ανταγωνιστική φορολογική πολιτική μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αποδεχόμαστε. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Η ελάχιστη φορολόγηση είναι μια λύση Ξέρετε ότι η όλη διαδικασία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει γοργά σε επίπεδο Συμβουλίου. Υπάρχει όμως κινητοποίηση της κοινή γνώμης. Υπάρχει και η διάθεση του Κοινοβουλίου να δράσει και σίγουρα του Επιτρόπου για τις Οικονομικές Υποθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το κοιτάξουμε λοιπόν και θα αναζητήσουμε λύσεις. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει όριο στο χρόνο ομιλίας. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να παραμένετε στο ένα λεπτό για τις ερωτήσεις και στο ένα λεπτό για την επερώτηση. Ε, ο κύριος Χωσέ Γκαρσία Μαργκάγιο Εμαρφίνη. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε, κύριε υποψήφια Επίτροπε. Μιλήσατε στην ε, ε, δήλωσή σας για επιβράδυνση οικονομική, αλλά κάποιοι πιστεύω ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας κρίσης. Όχι κρίση ζήτησης ε, σαν αυτή το Lehman Brothers, αλλά κρίση προσφοράς που οφείλεται σε, ε, στις, εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, τεχνολογικούς πολέμους, το Brexit, ε, η, η επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζετε ε, όλα, αυτά γιατί διτελέσετε και υπουργό Εξωτερικών. Χρειάζονται λοιπόν κάποια διαρθρωτικά μέτρα, αλλά με βάση ε, τη δηλώση κυρίας Λαγκάρτ που μοιάζει πολύ ε, με τον Τράγκη, ε, θέλει ελαστικοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής ε, και ενίσχυση της νομισματικής πολιτικής. Πώς όμως ε, με τόσο χαμηλά επιτόκια μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να επηρεάσουμε τη σταθερότητα των ε, τραπεζών. Επίσης μιλήσατε για κάποια ελαστικοποίηση. Οπότε σκέφτεστε να μην περιλάβετε όχι για στατιστικούς λόγους τις επενδύσεις σε κάποιους τομείς, οικολογική μετάβαση, βοήθεια προς κάποιους, κάποιες σημαντικές τεχνολογικές επιχειρήσεις τι πρέπει να προσθέσουμε στις πολιτικές που βέβαια είναι σαν να δίνουμε ασπιρίνη για να ε, θεραπεύσουμε τον καρκίνο και όχι ε, εφαρμόσουμε τα διαρθρωτικά μέτρα που χρειάζονται. Ε, well, thank, thank you. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαργκάγιο. Δεν θα απαντήσω ισπανικά. Προηγουμένως αναφέρθηκα στις προβλέψεις, τις ε, προβολές του Νοεμβρίου. Και ακριβώς γιατί το Ινστιτούτο αυτό έχει μεγάλο κύρος. Κοιτάζουν όλοι βεβαίως τις προβλέψεις διαφορετικών φορέων από όλο τον κόσμο, διαφορετικών Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων και ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρή επιβράδυνση. Αυτή η επιβράδυνση θα μπορούσε να έχει μια περισσότερο μακροχρόνια διάρκεια από ότι αναμέναμε πριν 6 μήνες ή ένα χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να επαφιόμεθα μόνον στην νομισματική πολιτική. Συζητούμε την νομισματική πολιτική και τις αποφάσεις της ΜΕΝ και δεν θέλω να σχολιάσω τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξορισμού δεν θέλω να αναλάβω τέτοιο σχολιασμό. Γνωρίζετε όμως, τουλάχιστον επ' αυτού πιστεύω όλοι συμφωνούμε, ότι από μόνη της η νομισματική πολιτική δεν εξαρκεί. Δεν εξαρκεί για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δυσχερής. Και μια ενδεχόμενη επιβράδυση διαρκείας στην ανάπτυξή μας. Δεν μιλώ για ύφεση, μιλώ απλώς για πολύ αργή, για ε, αργό ρυθμό στην ανάπτυξη. Τι θα πει αυτό. Περισσότερο συντονισμό θέλουμε στη δημοσιονομική πολιτική, επενδύσεις και διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Είναι νομίζω ενδιαφέρον να δούμε ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής για το ευρώ μια από τις αποφάσεις που ελήφθη αφορούσε ακριβώς αυτό το εργαλείο του προπολογισμού για την σύγκληση, τον ανταγωνισμό και με στόχο να δώσει περισσότερη όθηση στις διαδοτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Θα δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν και πώς θα προχωρήσουν. Όμως αυτός είναι ο στόχος και πάει στην κατεύθυνση που αναφέρατε. Επερώτηση υπάρχει. Δεν ξέρω τι ε, ονειρευτήκατε σήμερα το βράδυ, αλλά τρει φορέ μιλήσατε για 27 προπολογισμού, ενώ ακόμα είμαστε 28 κράτη-μέλη. Έγινε λόγο για φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, ε, τελωνία και για το Brexit για παράδειγμα. Το σύνορο Βορείου Ιρλανδίας Ιρλανδίας είναι μείζον πρόβλημα και είναι το προηγούμενο που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει η Βρετανική κυβέρνηση για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης θέλει να δημιουργήσει μια Σιγκαπούρη στην άλλη πλευρά της μάχης. Επίσης, ε, έγινε λόγος για φορολογικούς παραδείσους. Θέλω να είμαι συγκεκριμένη. Έχουμε ε, το Γιβραλτάρ στις πύλες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί δεν υπάρχει φόρος ε, πλούτου, δεν υπάρχει φόρος πολίσεων. ο φόρος στα τυχερά παιχνίδια είναι 0,5% και 10% είναι ο φόρος εταιριών και μάλιστα μόνο εφαρμόζεται σε καμία ουσιαστικά επιχείρηση. Οπότε έχει δημιουργήσει μια διαφορά εισοδήματο 1 προ 6 σε σχέση με το Γιβραλτάρ και την ε, υπηρετική ε, πλευρά. Οπότε, τι θα κάνουμε για τους φορολογικούς μας παραδείσους και τι πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να γίνει ώστε στις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουμε ένα ε, φορολογικό καθεστώς που ουσιαστικά θα είναι ε, ανύπαρκτο και θα δημιουργήσει τεράστιους κινδύνους για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους εθνικούς κορβανάδες. Ευχαριστώ. Ναι, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και ξεκάθαροι την ημέρα μετά της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί αυτόματα σε τρίτη χώρα. Δεν ήταν αυτό η επιθυμία μας, δεν ήταν αυτό το δικό μας σχέδιο, αλλά θα μπορούσε να είναι η αυτόνομη και κυρίαρχη απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Είδα το διάλογο του Πρόεδρου Ζαν Κλοντιούνκερ και του Βρετανού Πρωθυπουργού. Τι να πω για μας. Δύο πράγματα. Πρώτον, το Ιρλανδικό σύνορο δεν θα είναι σκληρό σύνορο. Θα πρέπει να σεβαστούμε πλήρως τι συμφωνίε της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη μετά τον Brexit στην Ιρλανδία. Δεύτερον, θυμάμαι τις δυσκολίες που είχαμε ε, με τη συμφωνία με την Πρωθυπουργό Μέη για το Γιβραλτάρ. Τότε είχαμε καταλήξει με κάποιο τρόπο ε, σε κάποια συμφωνία μεταξύ ε, της δικής της κυβέρνησης και της Βρετανικής κυβέρνησης και τώρα και το Ηνωμένο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τηρήσουν αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει πολύ περιοριστικό βασικό προσανατολισμό ε, στην δημοσιονομική πολιτική στις ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές της η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε ένα ε, πρόγραμμα βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη και οι επενδύσεις αυτές σίγουρα δεν θα είναι αποκλειστικά ιδιωτικές. Αντιθέτως, ο δημόσιος τομέας θα παίξει ρόλο κλειδί ε, για να αντισταθμίσει τις αποτυχίες ε, της αγοράς, για να έχουμε βιωσιμότητα και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και την αλλαγή του κλίματος. Συμφωνείτε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Green Deal, η κινητοποίηση ε, ιδιωτικών αλλά κυρίως δημοσίων επενδύσεων θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και ε, από εκεί θα πρέπει να έχουμε τον προσανατολισμό για το μέλλον και να εξετάσουμε τον προσανατολισμό που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σούστερ. Αυτή η πράσινη συμφωνία, το Green Deal, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν το κατέστησε αυτό απόλυτα σαφές. Προσωπικά συμφωνώ με αυτό. Ο αριθμός 1 τρισεκατομμύριο που ανέφερε η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό. Θα εργαστούμε σκληρά Προσωπικά θα συνεργαστώ με τους αντιπροέδρους Τίμερμανς και τον Πρόφσκης, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα για να κινητοποιήσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο προφανώς, για να πετύχουμε όμως έναν τέτοιο στόχο θα πρέπει να προσθέσουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιους πόρους. Θα πρέπει να έχουμε δημόσιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό, το σχέδιο επενδύσεων για τη βιώσιμη Ευρώπη, ξεκινάει παράλληλα με το πρόγραμμα Invest EU, το οποίο νομίζω ότι θα συμβάλλει σημαντικά στο σχέδιο επενδύσεων ε, λόγω των δυνατοτήτων που θα συγκεντρώσει το πρόγραμμα αυτό σε νέα προγράμματα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε σημαντική συμμετοχή κεφαλαίου. Στις εργασίες μας θα πρέπει να συνεχίσουμε και τις εργασίες πάνω στα πρότυπα για τα πράσινα, τα οικολογικά ομόλογα. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας στο εγγύς μέλλον και οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει όπως γνωρίζετε. Επερώτηση, ναι ευχαριστώ. Επιτυχής εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής επενδύσεων ιδιαίτερα αν πετύχουμε και την οικολογική μετάβαση στην οικονομία, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρώπης. Για να έχουμε δίκες ε, και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού, νομίζω ότι ε, είναι απαραίτητο αυτό που είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, να έχουμε έναν πράσινο... Θα πρέπει να έχουμε το Green Border Adjustment. Εσείς ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου προγράμματος. Όπως σας είπα, οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει εντός των υπηρεσιών μας και το μήνυμα είναι απόλυτα σαφές. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα επενδυτικών κεφαλαίων για επενδύσεις με συγκεκριμένο στόχο και ιδιαίτερα με περιβαλλοντικό στόχο. Θέλουμε λοιπόν ε, με τα πράσινα ομόλογα να θέσουμε ένα σημείο αναφοράς στις αγορές και νομίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε ένα πολύ θετικό επενδυτικό κλίμα από πλευρά των επενδυτών. Δεν θα μπορούσε η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να λείπει στον τομέα αυτόν. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μείνει πίσω ένα τέταρτο. Παρακαλώ λοιπόν να, να τηρείτε στο μέλλον το χρόνο σας. Ο Ζιλ Μποαγέ από το Renew Europe. Oui, merci, monsieur le commissaire désigné. Alors, pendant... Σας ευχαριστώ. Κύριε υποψήφια, κύριε υποψήφια επίτροπε, στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία ε, εξεπλάγην που οι πολίτε με ρωτούσαν για το θέμα τη φορολογική εναρμόνιση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το θεωρούσα τεχνικό θέμα, αλλά ανακαλύπτω ότι είναι πολιτικό θέμα που μάλιστα απασχολεί ιδιαίτερα του Ευρωπαίου πολίτε. Και αυτό φάνηκε και από τι ερωτήσει των συναδέλφων και όχι μόνο των Γάλλων. Οπότε, σας ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δυστυχώ η ε, αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών, λόγω κυρίω τη διαδικασία ε, τη ε, ομοφωνία στην ψηφοφορία. Και μάλιστα χρειάζεται ομοφωνία για να καταργηθεί ο κανόνα τη ομοφωνία. Κάτι που είναι παράδοξο. Ούτε και εμεί έχουμε ομοφωνία βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η πλειοψηφία θέλει στην συγκεκριμένη κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε απτή πρόοδο και φυσικά δεν μπορούμε τέτοια περίπλοκα προβλήματα να τα λύνουμε μία νυχτή, αλλά θα πρέπει να ε, διαχωρίσουμε το πρόβλημα αυτό, να το επιμερίσουμε σε μικρά σταδιακά βήματα. Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο μέτρο, η πρώτη δράση που θα μπορούσατε να μας προτείνετε ώστε αυτή η θητεία στην οποία ελπίζω να συμπορευτούμε ε, θα μπορούσε να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ κύριε Μπόγε. Όπως είπατε κι εσείς, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση για την κατάργηση της ομοφωνίας, του κανόνα της ομοφωνίας στην ψηφοφορία. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο. Και όχι από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αλλά, όπως είπα και στην αρχική μου δήλωση, θα χρειαστούν τεράστιες πολιτικές προσπάθειες. Και μόνο η πολιτική εμ, υποστηρίζοντας την κοινή γνώμη ε, τους ενδιαφερομένους, τους ενεχομένους και μία ευαισθητοποίηση από τις χώρες που έχουν διαφορετική γνώμη θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο. Το άρθρο 116 είναι λίγο διαφορετικό, γιατί προβλέπει ότι υπό συγκεκριμένου νομικούς όρους και προϋποθέσεις θα ήταν, αν όχι πιο εύκολο, τουλάχιστον πιο σαφές. Αλλά στην ρήτρα Πασρέλ Απαιτείται τεράστια πολιτική προσπάθεια. Και θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Και θα είναι από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα αναλάβω. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να μην εφαρμόσει το ψηφιακό φόρο. Οι τρεις χώρες που δεν συμφωνούσαν είπαν ότι δεν διαφωνούσαν γενικώ, αλλά ήθελαν να περιμένουν να αναπτυχθεί μια συνένεση παγκοσμίω. Και αυτό θα το δούμε στο μέλλον, τους επόμενους μήνες. Και θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό το 2020 και ίσως αναθεωρήσουμε θέση. Παρακαλώ, μισό λεπτό για την επερώτηση. Καλώς. Αναφερθήκατε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ε, G20, ΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ισχυρή στις διαπραγματεύσεις αυτές μόνο αν έχει ενιαίο μέτωπο. Δηλαδή αν έχουν προηγηθεί κάποιες κοινέ θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί θα παρακολουθούμε είναι και σε αυτά τα θέματα και θα επαγρυπνούμε στο μέτρο. Ελπίζω κι εσείς το ίδιο να επαγρυπνείτε και μετα... αφού αναλάβετε τα καθήκοντά Τα καθήκοντά και η κυρία Φόντερ Λάιν επίσης. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολλές, πολλές πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες στη συζήτηση στον ΟΣΑ. Πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες τώρα από ότι λίγους μήνες πριν. Δεν είμαι υπεραισιόδοξος, αλλά σίγουρα είμαι λιγότερο απεσιόδοξο σήμερα από ό,τι πριν από μερικούς μήνες. Γιατί οι συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ έχουν οριμάσει κάπως, έχουν προχωρήσει και υπάρχει δυνατότητα να βρει λύσεις. Ευχαριστώ. Ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες, έχει το λόγο από την Επιτροπή Απασχόληση και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ορισθέντα Βίτροπε, σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τις αρνητικές επιπτώσεις της, τα σοκ ε, εσωτερικό στην αγορά των κρατών μελών. Μιλήσατε για ένα πρόγραμμα αντασφάλιστης για την ανεργία, παροχών ανεργίας. Είναι φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα. Όμως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς η θέση σας το πρόγραμμα αυτό θα είναι επιδόματα ή θα είναι δανειοδότηση προς τα κράτη-μέλη ή ένα μείγμα και των δύο. Και έπειτα θα προβλέπετε για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνο για τα κράτη της Ευρωζώνης. Και ακόμα ε, επιπλέον τι θα απαιτείτε για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη αυτά να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την αντασφάλιση, αυτό το πρόγραμμα αντασφάλισης για την ενεργεία. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Η αρμοδιότητα που μονατέθη στην επιστολή αρμοδιοτήτων ορίζει ακριβώς και τα του προγράμματος. Οπότε πρόκειται για μια αρμοδιότητα, για μια αποστολή που δεν θα ολοκληρωθεί εδώ κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Δεν είναι και τόσο απλό. Υπογραμμίσατε τα βασικά στοιχεία ούτω ή άλλω του προγράμματο με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και έχω ήδη ε, πει ότι αυτό το εργαλείο δεν θα πρέπει να είναι κάποια πράγματα, όχι μόνιμες μεταφορές, όχι αποδυνάμωση των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, όχι ένας αυτόματος μηχανισμός εκταμίευσης. Θα συζητήσουμε διεξοδικά τα δύο-τρία σημεία τα οποία απαριθμίσατε. Δάνεια στήριξη στον προπολογισμό. Θα το δούμε. Προφανώς, σε τέτοιες συνθήκες, ανάλογα με την ε, αγορά, τα δάνεια είναι ένα εργαλείο κάπως πιο αδύναμο, με λιγότερη ε, επίδραση από ότι η άμεση υποστήριξη του προπολογισμού. Όμω η στήριξη του προπολογισμού απαιτεί και πολλά, πολλά ποσά, μεγάλα ποσά. Διότι αν υπάρξουν εξωτερικοί τριγμοί, εξωτερικά σοκ, και μάλιστα ταυτόχρονα σε πολλά κράτη, η στήριξη προς τον προπολογισμό χωρίς σοβαρή μεγάλη χρηματοδότηση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τα μελετάμε όμως και στον ορισμό θα δούμε τι επιτρέπεται να προβλέψουμε ως δυνατότητα. Ένα, αρχικό, ένα πρόγραμμα από την αρχή να είναι σύστημα δανειοδότησης και σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς την άμεση υποστήριξη του υποπολογισμού. Θα το δούμε. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι τι επόμενε εβδομάδες, διότι έχω αναλάβει τον ορισμό αυτό να τον ε, ολοκληρώσω τάχιστα, θα είμαστε μαζί στην προσπάθεια. Η ερώτηση όμως ήταν θα ακολουθήσετε την κοινωτική μέθοδο για, την, ε, για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σύστημα αντασφάλισης για την ενεργεία. Διότι σε αυτή την περίπτωση, εάν πρόκειται για δάνεια, θα πρέπει να υπάρχει κάποια εγγύηση σχετικά εντό του προπολογισμού. Τι ποσό πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει αυτή η εγγύηση. Εάν τώρα πρόκειται για επιδοτήσεις, πάλι θα πρέπει να τους αναλογεί κάποιο ποσό. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτό το χρηματικό ποσό έχει οριστεί ή τέλος πάντων τα όρια του, ανώτατα και κατώτατα. Άρα, <clears throat> απαντήσατε κι εσείς στις ερωτήσεις σας. Διότι αυτό που πρέπει να καθορίσουμε υπονοεί ότι στην περίπτωση ενός προγράμματος δανείων ή άμεσης υποστήριξης τον προπολογισμό, οι συνέπειες θα είναι δυο λογιών διαφορετικές. Στην πρώτη περίπτωση, οι συνέπειες αυτές είναι σχετικώς εύκολες να τις χειριστούμε. Στις άμεσες μεταφορές προς τον προπολογισμό και πάλι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ότι θα πρέπει κάπως να θεμελιώνονται σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε λίγες εβδομάδες ναι. πιστεύω όλα αυτά θα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα έχουμε τον ορισμό του προγράμματος ε, και θα δούμε τι συνέπειες θα φέρουν οι μέθοδοί μας στις κοινοτικές μας αποφάσεις. Ευχαριστώ, Ήρωη Ναλόμα από το S&D. Κύριε Τζεντιλόνι, έχετε πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό και νομίζω ότι όλα τα προσόντα σας θα είναι πλεονέκτημα στα ε, στο δύσκολο έργο που σας περιμένει. Όσον αφορά την ε, φορολογία των εταιριών ε, και με έχουν πάρει διάφοροι τηλέφωνα, μου έχουν πει ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει περισσότερο όσον αφορά τη φορολογία των, τη φορολογήση των εταιριών. Χρειάζεται και ψηφιακός φόρος, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μπορείτε να μας περιγράψετε τις βασικές σας προτεραιότητες κατά τη φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών και ιδιαίτερα ε, των ε, ψηφιακών εταιριών και πώς βλέπετε το ρόλο σας στις συνεχιζόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις για την ψηφιακή φορολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαϊναλούμα. Ο στόχος νομίζω είναι σαφής. Η ψηφιακή επανάσταση πρώτη φορά μας έφερε σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση όπου δημιουργείται αξία συχνά και μέσω των προσωπικών μας δεδομένων. Οι φόροι όμως δεν καταλήγουν στον ίδιο τόπο όπου παράγεται η αξία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και εγώ πιστεύω το εξή. Μετά από διάφορε κάποιε αρχικέ δυσκολίε ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά τα αποτελέσματα τη ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίσαμε να κρατήσουμε τα καλύτερα στοιχεία από τη διεθνή συζήτηση στον ΟΣΑ, παράδειγμα. Και μπορεί αυτό να φαίνεται σαν στρατηγική εξόδου από δυσκολίες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα υπάρχει πραγματική ανησυχία, ιδιαίτερα από πλευράς των Ηνωμένων ε, Πολιτειών, και υπάρχει διάθεση να βρεθούν λύσεις, να βρεθεί συμβιβασμός στον ΩΣΑ. Η Ευρώπη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να βρούμε του χρόνου λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Επερώτηση. Ναι, κύριε Τζεντιλόνη, στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε ότι εάν δεν υπάρξει διεθνής συμφωνία θα υποβάλλεται ευρωπαϊκή πρόταση για ψηφιακό φόρο. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε αποτελέσματα είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε ως πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη του χρόνου, εντό του 2020. Ναι, το πρόγραμμά μου, το χρονοδιάγραμμά μου είναι σαφές. Εάν δεν υπάρξει συνένεση του χρόνου σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρξει η ευρωπαϊκή πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι το τρίτο τρίμηνο του χρόνου θα ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή πρόταση. Δεν θα βιαστούμε να εκπονήσουμε ευρωπαϊκή πρόταση κατά τη διάρκεια της ε, διεθνούς συζήτησης, της ε, συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεσμεύομαι όμως σοβαρά, δεσμεύω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουμε πρόταση του χρόνου, εφόσον δεν δημιουργηθεί συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος Έρνστ Ουρτασούν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνι, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας οικονομικής επιβράδυνσης και ως Επίτροπος Οικονομίας θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε και μάλιστα χωρίς να έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς σταθεροποίηση και με κανόνες που έχουν ε, προκαλέσει μεγάλα ασφάλματα της ευρωπαϊκής πολιτικής στο παρελθόν και υπάρχει κίνδυνος επανάληψη αυτών των λαθών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και ήδη είπατε ότι θα γίνει η αναθεώρηση και του εξάπτυχου και του δίπτυχου πακέτου και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά ε, θα ήθελα να μου πείτε, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είπε ότι οι κανόνες μας έχουν ένα προκυκλικό χαρακτήρα. Και μάλιστα ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε το ίδιο πράγμα. Εσείς συμφωνείτε ότι οι παρόσες ε, διατάξεις έχουν αυτή την προκυκλική ε, κατεύθυνση και τι πιστεύετε ότι πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αποφύγουμε αυτό το προκυκλικό χαρακτήρα και την το προκυκλικό αποτέλεσμα του εξάπτυχου και δίπτυχου πακέτου στη μεταρρύθμιση. Ναι, ο κίνδυνος του προκυκλικού αποτελέσματος είναι εμφανής και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ήδη επισήμανε αυτόν τον κίνδυνο και μάλιστα πολύ ξεκάθαρα. Και αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε κατά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου των, των δύο δεσμομέτρων, του εξάπτυχου δηλαδή και του δίπτυχου πακέτου, είναι τι μέλη γενέστε. Εγώ προσωπικά εκτιμώ τη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να είναι απλά τα μέτρα ε, εύχριστα, να εφαρμόζονται εύκολα και να είναι αντικυκλικά. Και αυτή η φιλοσοφία και αυτή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη και κάποιες αντιρρήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Να μην είναι δηλαδή υπερβολικά περίπλοκα τα μέτρα, να μην αφήνουν ε, μεγάλο περιθώριο λιγμών, όπως είναι οι σημερινοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πάντως, η απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε, ποια θα είναι η μελλοντική μας πορεία μετά την αξιολόγηση του εξάπτυχου και δίπτυχου, ε, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα είναι διόλου εύκολη αυτή η απόφαση. Εγώ ε, τονίζω πάντα την ε, φιλοδοξία και θα ήθελα να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες, να είναι πιο αντικυκλικοί και να εφαρμόζονται πιο εύκολα. Πάντως, σέβομαι και τη γνώμη που λέει προσοχή, σύνεση, γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε τα ίδια προβλήματα με κάποια μέσα εργαλεία ε, ερμηνείας χωρίς να ανοίγουμε τη δυνατότητα για κάποιες νομοθετικές αλλαγές. Πάντως όλα αυτά θα αποφασιστούν πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους. Επερώτησε ο κύριος Φορτασούν ένα μεγάλο τμήμα θα, ε, το, θα, θα αναλάβετε εσείς για να δώσετε τις βασικές κατευθύνσεις των αλλαγών. Εσείς είστε επιφορτισμένος με αυτό το θέμα. Επίσης, υπάρχει η διαδικασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών, που πολύ έξυπνα το αναφέρετε στις γραπτές απαντήσεις. Στο παρελθόν είχαμε μια αναποτελεσματική και όχι συμμετρική ε, εφαρμογή της διαδικασίας των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πώς πιστεύετε ότι αυτό το μέσο ε, μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Επίσης, ε, μιλήσατε για τους κινδύνους αγοράς ακινήτων σε αυτές τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις ιδέες σας. Πώς θα διορθωθούν αυτές, πώς θα χρησιμοποιηθεί το μέτρο για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η ανάλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ήταν πολύ χρήσιμη γιατί έδωσε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατημέλη κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες ιδέες, προτάσεις όχι μόνο για τα κλασικά χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και για άλλα ζητήματα. Το ιδιωτικό χρέος, την αγορά των ακινήτων, την κατάσταση στην υγεία. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες. Και οι καταστάσεις αυτές ε, και γι' αυτό θα πρέπει στο μέλλον να τις ενισχύσουμε. Η Φραντζέσκα Ντονάτο από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Κύριε Τζεντιλόνη, στις γραπτές σας απαντήσεις σας στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου δεσμεύεστε να προβλέψετε μια πολιτική ατζέντα για τη στήριξη της ανάπτυξης, βρίσκοντα τη σωστή ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας και τη λύση κάθε προβλήματος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, με ευελιξία εντός των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ερωτώ, τι εννοείται με τη δέουσα ευελιξία. Ποιε είναι οι παράμετροι που θα εγκρίνετε και οι μεταβλητέ που θα λάβετε υπόψη για να αποφασίσετε εάν θα παρέχετε περισσότερη ευελιξία ή όχι στη διαχείριση του προπολογισμού του σε ένα κράτο μέλο ή όχι. Ε, είναι πολιτική εντελώ η απόφαση. Θα δίνετε ευελιξία στι κυβερνήσει που είναι ε, φιλικέ προ εσά, που σα είναι συμπαθεί, ή θα χρησιμοποιείτε κριτήρια αξιολόγηση που θα λαμβάνουν πραγματικά υπόψη τι προοπτικέ ανάπτυξη και τι ανάγκε για επενδύσει των επιμέρου κρατών μελών. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Ντονάτο. Η ευελιξία αυτή πρόκειται και σε κανόνες. Κανόνες που ορίζονται από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτούς που επικαιροποίησαν το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι βασικές παράμετροι. μέσω του διαλόγου που είναι άκρο αναγκαίο ε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυβερνήσεων κρατών μελών. Έτσι ορίζονται τα όρια τη ευελιξία. Ο διάλογο αυτό, αυτή η γραμμή δράσης είναι απαραίτητη και τα προγράμματα που υποβάλλονται από τις κυβερνήσεις αφορούν κυρίως τις επενδύσεις. Υπάρχει ρήτρα πολύ συγκεκριμένη για τις επενδύσεις. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Οι έκτακτες ε, περιστάσεις λαμβάνονται σαφώς υπόψη. Μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίζει πρόβλεπτα γεγονότα έκτακτου χαρακτήρα δεν πιστεύω ότι στην αξιολόγηση, στη θεώρηση αυτή της, αυτής της ευελιξίας, αυτής της ελαστικότητας, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική επιλογή και διακριτική μεταχείριση, ε, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς πολιτικός έχετε διαφορετική άποψη, αλλά σε ό,τι με αφορά το κριτήριο της ελαστικότητας, της ευελιξίας, θα πρέπει να βασίζεται στις κατευθύνσεις και στα όρια που ορίζει το σύστημά μας. Επερώτηση. Όμως, για να ανακάμψει, για να τονωθεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, είπατε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε εκτατικές δημοσιονομικέ πολιτικέ και να υπάρχει παραγωγική κρατική δαπάνη. Όμω, χώρε με μεγάλο δημόσιο χρέο όπω η Ιταλία καλούνται να είναι προσεκτικέ, ώστε να μείνουν στα όρια του δημοσιονομικού χρέου που ορίνει, ορίζει το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Δεν γίνεται όμω έτσι να γίνουν και επενδύσει στι πιο καθυστερημένε περιοχέ, όπω το νότο τη Ιταλία και στα νησιά. Άρα, πώ θα μπορέσετε ε, να προωθήσετε τον χρυσό κανόνα για τις επενδύσεις και για τις υποδομές, την έρευνα, για την ε, οικολογική ε, χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία και πώς τελικά θα μπορεί αυτό να αφαιρεθεί από τον κρατικό προπολογισμό εφόσον θα έχει τέτοιο στόχο το σκέλος των επενδύσεων. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, ήδη σήμερα Γίνεται διάλογος στα πλαίσια του εξαμήνου με τις επιμέρους κυβερνήσεις. Και με τη ρήτρα των επενδύσεων προβλέπεται αυτή η εφαρμογή η χρήση μεγαλύτερων περιθωρίων ελαστικότητας και ευελιξίας σε χώρας με τέτοιο προπολογισμό. Συζητάτε το αν θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε τον χρυσό κανόνα. Λόγω χάρη στη γνωμοδότηση του Ταμείου, του, συγγνώμη, του Συμβουλίου, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τις κρατικές επενδύσεις, εφόσον ε, συνδεθούν, σχετιστούν απευθείας με περιβαλλοντικούς στόχους. Είναι ένα θέμα σοβαρότατο που θα συζητηθεί τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστούμε ο κύριος Φίτο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να πω, να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα εάν θεωρείτε σκόπιμο, θετικό, να παρέμβετε για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με ένα από τα βασικά στοιχεία του προπολογισμού, τους πόρους, που προβλέπονται για τα επιμέρους ε, κράτη, συγγνώμη, και μιλώ για τα ταμεία συνοχής. Η πρόεδρος της Επιτροπής έχει ανακοινώσει πολλά σημαντικά προγράμματα για την ανάπτυξη και την οικονομική αύξηση και μίλησε και για ενδεχόμενη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ω προ την αναθεώρηση λοιπόν αυτή, θα σα ρωτώ το εξή συγκεκριμένο. Μπορείτε να μα πείτε χειροπιαστά το πώς μπορεί να υπολογιστεί η ποσόστο, το ποσοστό χρημα... συγχρηματοδότησης που προβλέπεται για τις επιμέρους χώρες στα πλαίσια του Ταμείου Σταθερότητας και σε σχέση με τις επενδύσεις. Διότι από τη μια φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάθεση να εξοδευτούν κάποια ποσά και μετά οι, επενδυσει αυτε επενδύσεις συνυπολογίζονται ξανά στο Σύμφωνο Σταθερότητα και αναπτυξη Είναι μια αντίφαση αυτό. Μπορείτε λοιπόν να μα πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό το θέμα διότι αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Κύριε Φίτο, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ερώτηση. Αλλά το θεμητόν του αιτήματο δεν χωρεί συζήτηση. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συζητιέται μάλιστα εδώ και καιρό. Απλώς και χρησιμοποιώ ως αφορμή την παρέμβασή σας για να πάω λίγο παραπέρα στο θέμα αυτό. Σε έναν κίνδυνο που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να διατρέξουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Δηλαδή, την υπόθεση, η διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων μας, που τώρα συζητούμε, το review, του εξαπτύχου και του διπτύχου μέτρων, του Σίξπακ και του ΤΟΥΠΑΚ, δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι θα λύσουν ταυτόχρονα όλα τα ζητήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην πολιτική μας ατζέντα, αλλά πολλές φορές είναι αντικείμενο διαφορετικών απόψεων ή διαφωνιών μεταξύ πολιτικών οικογενειών ή κάποιες φορές και μεταξύ χωρών. Δεν λέω λοιπόν ότι είμαι αντίθετο με αυτή την προοπτική, Απλώς οι κανόνες μας για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εξαρτηθούν από το τι θα αποφασίσουμε, ε, δηλαδή αν θα, τις, θα τους αλλάξουμε σε νομοθετικό επίπεδο, θέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά όχι να γίνει σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από το οποίο αφαιρούμε όλα του τα στολίδια και τελικά δεν μένει τίποτα. Ε, δηλαδή, επενδύσεις, περιβάλλον, αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Το, σύστημα το θέμα της συνοχής δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Δηλαδή, εφόσον μου θέτεται αυτό το ερώτημα, πρέπει να πω ότι Ακόμα πιο πολύ θα πρέπει να επαφιόμαστε στους νομοθετικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χρειάζεται δηλαδή μια σαφέστερη ερμηνεία πολλών από τους στόχους. Μάλλον, εάν δεν υπάρξει μια τέτοια ερμηνεία, δεν θα γίνεται και ρεαλιστικά τίποτα, εφόσον ε, πέρα από το πλαίσιο το στενά νομοθετικό. Ναι, αλλά στα πλαίσια του ίδιου συλλογισμού και βάσει των παρεμβάσεων που ακούσατε σήμερα σε σχέση με τους διαφόρους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των επιμέρους κρατών. Σας ερωτώ, δεν θεωρείτε ότι θα ήταν πολύ σκοπιμότερο και προσφορότερο σε καιρούς ευελιξίας να παρέμβει κανείς ώστε να αποφύγει σε επιμέρους χώρες ε, να υπάρχει ευελιξία ε, να υπάρχει ευελιξία που επιτρέπει μεγαλύτερε δημόσιε δαπάνε χωρί κανένα τελικό σκοπό. Χωρί να εξυπηρετούν κανένα τελικό σκοπό. Θα έπρεπε η ευελιξία ενδεχομένω να συνδεθεί απευθεία με τι επενδύσει, συνδεόμενη ε, και προβλέποντα ένα τέτοιο κανόνα στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Διότι σε κάποιε χώρε θα αντιμετωπίσουμε την περίπτωση προτάσεων όπου θα έχουμε περισσότερε δημόσιε δαπάνε τη ευελιξία, χωρί να γίνονται δημόσιε επενδύσει και τελικά θα περάσουμε σε στρεβλού δημοσιονομικού κανόνε που θα δημιουργούν αστάθεια στην Ευρωζώνη μακροπρόθεσμα. Ναι, πρέπει να επικεντρωθούμε στι επενδύσεις, στι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. αυτό που κάνει να αναπτυχθούν οι οικονομίε μα. Αν δούμε του προπολογισμού των τελευταίων ετών. Με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη επέτρεψε να αποφύγουμε μεγαλύτερε ε, κρίσει, χειρότερε κρίσει. Ήταν καλό για τη μείωση του χρέου, αλλά δεν μπόρεσε να περιορίσει αποτελεσματικά το χρέος. και δεν μπόρεσε να βελτιώσει την ε, ανάπτυξη και τις επενδύσεις μέσω των διευθυντικών ταμείων. Γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας αυτούς τους στόχους στα πλαίσια της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. κύριος Μουρεζάν από την Επιτροπή Προπολογισμών ΕΛΚ. Thank Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ορισθέντα Επίτροπε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σα τον αντίκτυπο των αποφάσεών σα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι σαφέ ότι μετά τον Brexit θα χρειαστούμε επιπλέον πόρου για να χρηματοδοτήσουμε τι παρούσε και τι νέε προτεραιότητέ μα. Και γι' αυτό η συζήτηση σχετικά με του ίδιου πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντική από ποτέ την εφαρμογή ε, του συνοριακού φόρου άνθρακα ε, Πιστεύετε ότι αυτός ο φόρος θα ενσωματωθεί στο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει στο παρελθόν να ε, τροποποιήσει το σύστημα ιδίων πόρων. Τι ε, θα κάνετε διαφορετικά διότι τώρα ή ποτέ πρέπει να πετύχετε. Και η τρίτη μου ερώτηση αφορά το συνοριακό φόρο άνθρακα. Πώς θα τον εφαρμόσετε για να μην επηρεάσετε αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Όσον αφορά τους ίδιους σπόρους, πράγματι, πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό μου. Δεν είναι δική μου δηλαδή. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου, δεν τις ακούσαμε. Δύο πράγματα λοιπόν. Πρώτον, Οι δασμοί της Τελωνιακής Ένωσης ε, είναι θεμελιώδους σημασίας για το σύστημα ιδίων πόρων. Γίνεται συζήτηση σχετικά με το ποσοστό του 10 ή του 20% που θα πρέπει να ανήκει στα κράτη-μέλη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για το ΦΠΑ. Δεν βλέπω να υπάρξουν άμεσες συνέπειες των αποφάσεών μας ε, στο ΦΠΑ ή στους νέους πόρους. Όσον αφορά τα νέα εργαλεία που σχετίζονται με τους νέους πόρους, οι πιθανοί νέοι πόροι από τη φορολόγηση και από το συνοριακό φόρο, άνθρακα δηλαδή, και την ε, κοινή φορολογική βάση των εταιριών. Και τα δύο αυτά είναι θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σοβαρά. Αν θέλουμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας ήδη κατά την ε, αρχή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Διότι δεν νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα μπορούμε να έχουμε κάτι ήδη μέσα στους επόμενους μήνες. Σε συνεργασία λοιπόν με την Επιτροπή σας, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε γρήγορα και αποτελεσματικά πάνω στον συνοριακό φόρο άνθρακα, αλλά οι νομικές και τεχνικές πτυχές δεν είναι εύκολο να καθοριστούν, όπως γνωρίζετε. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα όλες αυτές τις δυσκολίες, γι' αυτό λέω ότι τώρα χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο και χρειαζόμαστε έναν επίτροπο ικανό να πείσει τα κράτη-μέλη και εσείς είστε πρώην υπουργό. Μιλήσατε για το ε, χαρτοφυλάκιό σας, ε, γι' αυτό σκέφτομαι τις μετοχές ε, και την ε, Amazon. ο ψηφιακός πόρος θα ενταχθεί στους ίδιους πόρους, η πρώτη μου ερώτηση και δεύτερον τι μέγεθος προβλέπετε για τους ίδιους πόρους ε, ε, στον επόμενο προϋπολογισμό. Και είσαστε επίτροπος για την οικονομία, όχι για ε, το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό θα ήθελα συγκεκριμένη απάντηση. Θέλω να έχουμε πιο ισχυρή βάση ίδιων πόρων διότι προϋπολογισμός που να βασίζεται μόνο στο ΑΕΠ Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα, είναι μάλλον αναπόφευκτο, αλλά δεν αρκεί για την Ένωση και το μέλλον μας. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους ίδιους πόρους. Η προηγούμενη Επιτροπή υπέδειξε τρεις τρόπους να ενισχύσουμε τους ίδιους πόρους και εγώ θα ασχοληθώ με αυτούς που εμπίπτουν στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, με όλη την πολιτική δύναμη και αποφασιστικότητά μου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω περί αυτού. Now, Engin Eroglu from... Ο Engin Eroglu από το Renew Αξιότιμε κύριε Τζεντιλόνι, για πολλούς πολίτες αλλά και για μένα ε, είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ε, όποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες του είναι ελεύθερος και όποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ε, για τις, τις πράξεις του ε, αναλαμβάνει και την ευθύνη για την δαπάνη των ε, μέσων του. Ε, αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε έχουμε ηθικό κίνδυνο και ασυμμετρία. Το ίδιο συμβαίνει εντό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσεις και ευθύνε πρέπει να βρίσκονται στα ίδια χέρια και πρέπει να δαπανούμε με οικονομία τα, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πρέπει Γι' αυτό έχουμε την αρχή του no bail, της ε, μη διάσωσης, ε, την έχουμε και στην ε, συνθήκη του Μάστριχτ. Εσείς σκοπεύετε να τηρήσετε την αρχή αυτή. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα την, το πρώτο μέρος της ερώτησή σας, διότι άργησα να βάλω τα ακουστικά. Τα δύο τρίτα άκουσα, δεν άκουσα την αρχή της παρέμβασής σας. Στο πρώτο τρίτο απλά ανέφερα ότι για πολλούς πολίτες και για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντική η ίδια ευθύνη, η οποία συνδέεται και με την ε, οικονομική χρήση των πόρων ε, και γι' αυτό ε, έθεσα και την ερώτηση σχετικά με την αρχή του no bailout. Uh, yes, it is a, a principle. Ναι, όντως. Συμφωνούμε με αυτή την αρχή και θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την αρχή της συλλογικής ευθύνης, κοινή ευθύνη. Και αυτό θα κάνω αν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Επερώτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγική σας ομιλία και χάρηκα που αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος ε, στο, στη φορολογία ε, και για περιβαλλοντικούς σκοπούς αλλά και τον ψηφιακό φόρο. Ε, οι προλαλήσαντες το ανέφεραν και δίνετε την εντύπωση ότι είσαστε προσιλωμένος στην εξέβρεση λύσης για τον ψηφιακό φόρο. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε ε, με σαφήνεια πού θα πάνε αυτοί οι νέοι φόροι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θα δαπανώνται ή θα υπάρχει κλίδα κατανομής στα εθνικά κράτη. Μα ναι, αλλά θα υπάρχει δέσμευση διεθνής. Με συγχωρείτε. Θα τα πω αγγλικά. Ήταν αυθόρμητη η αντίδρασή μου. Το να απαντήσω στα Ιταλικά. Θέλουμε λοιπόν ε, παγκόσμια δέσμευση όσον αφορά την ε, ψηφιακή φορολογία. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε αποτελέσματα κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι πριν κάποιους μήνες. Οι εξελίξεις ε, της συζήτησης στο πλαίσιο του ΩΣΑ κινείται μάλλον προς μια γενική φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων όχι μόνο δηλαδή τις ψηφιακές ε, πλατφόρμες, ε, αλλά όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, διότι ψηφιοποίηση βλέπουμε σε όλες τις πολυεθνικές ε, και όχι μόνο τις πολυεθνικές του ψηφιακού τομέα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δεχτεί η Ευρώπη. Ευχαριστούμε, Νικόλα εδώ είμαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, υποψήφια Επιτροπή. Διάβασα ότι μεταξύ των νομοδιοτήτων που σας αποδόθηκαν από την ε, πρόεδρο Φόντεν Λάιεν, δεν θα επανέλθω στι επενδύσεις, τις πράσινε επενδύσεις, λέει ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε να επιτύχετε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξη στο πλαίσιο των ε, βιώσιμων επενδύξεων και ότι θα κοιτάξετε βεβαίω να ισχύουν και να εφαρμόζονται κανόνε του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ε, το είπαμε επανειλημμένο σήμερα. Πώ πρόκειται όμω να απελευθερώσετε, να ενεργοποιήσετε αυτέ τι πράσινε επενδύσει σε χώρε με μεγάλο δημόσιο χρέο που δεν έχουν περιθώριο δαπανών. Διότι από την δική μα την οπτική γωνία δεν έχει νόημα να καταπολεμούμε τι κλιματικέ αλλαγέ, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει, ε, εφαρμόζοντα ίδια μέτρα και σταθμά για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν θα είχε λογική. Όταν λοιπόν λέμε ε, ανάγκε ε, δαπανών. Για να γίνει αυτό χρειάζεται τόλμη για να αρχίσουν να συζητώνται οι πολιτικέ λιτότητα που εφαρμόζονται τώρα. Και κοιτάζοντα λίγο το ιστορικό και την ε, πορεία σας, πάντοτε υποστηρίζατε και ε, στηρίζατε αυτές τις πολιτικές λιτότητα που κατά τη δική μα την άποψη οδήγησαν σε μια πραγματική κρίση και σε ύφεση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε κάθε περίπτωση έφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατάσταση με βαθύτερες ανισότητες κοινωνικές και οικονομικές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό των ε, κρατών. Τι σκέφτεστε να κάνετε από αυτού. Θα αμφισβητήσετε τις ε, πολιτικές της λιτότητας. Σας ευχαριστώ κύριε Πεντιτσίνη. όταν λέτε για τους κανόνες μας και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, και ότι δεν κατάφεραν αρκετά να επιτρέψουν την αύξηση των επενδύσεων, την, ε, ε, τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις να τις ευνοήσουν και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Εκεί φαίνονται και τα όρια των κανόνων μας, ε, παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι έχουμε και κάποια θετικά αποτελέσματα, κάποιες επιτυχίες, μείωση του ελλείμματος ή την ε, αποφυγή περαιτέρω σοβαρών κρίσεων. Αν το πούμε αυτό και το δούμε ε, σοβαρά. Δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, να, παραγνωρίζουμε τα εξή δύο. Ε, πρώτον, ότι σε κάθε περίπτωση οι κανόνες μας, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ήδη προέβλεπαν την δυνατότητα να δοθούν κίνητρα για δημόσιες και κρατικές επενδύσεις. Η περίφημη αυτή ε, ευελιξία για τις επενδύσεις, η ελαστικότητα προβλέπεται στους κανόνες μας. Και κατά δεύτερον, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη δική μας ε, χώρα προέλευσης που είναι η ίδια, ε, δεν θα πρέπει τη δυσκολία να προωθηθούν οι δημόσιες, οι κρατικέ επενδύσεις, να την αποδίδουμε πάντοτε στην ε, εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Υπάρχουν δυσχέρειε και δυσκολίε όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες εσωτερικώς ε, για την προώθηση των επενδύσεων. Ο ρυθμό προς τις επενδύσεις, η όθηση και αυτός ο αγώνας, ε, αυτό ο διαγωνισμό για να γίνουν καλύτερες επενδύσεις. Λείπουν οι πόροι και δεν φταίει μόνο η Ευρώπη γι' αυτό. 10 δευτερόλεπτα μόνον για επερώτηση. Απλώς να πω ότι αν μου επιτρέπετε, η Ιταλία έχει μπλοκαριστεί, επειδή αναφέρατε την Ιταλία, έχει μπλοκαριστεί από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αλλά και ιταλικό ταυτόχρονα που περιορίζει τις επιπτώσεις του δημόσιου χρέους με ε, πραγματικές ε, επιπτώσεις να εμποδίζονται οι κρατικές επενδύσεις. Εάν μπορούσαμε να παρέμβουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να μην ε, μπορούμε να παρέμβουμε στις πρωτογενείς αγορές, ίσως θα απελευθερώνταν τεράστια ποσά για χώρες όπω ε, όπως η Ιταλία που έχουν μεγάλη πρόοδο οικονομική, πρωτογενέ, δηλαδή πλέον κάθε χρόνο, αλλά δεν μπορούν να τα επενδύσουν. Δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ναι, Κοιτάξτε, σέβομαι την άποψή σας, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που ε, είναι το καθήκον μας ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Να γίνουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότεροι για την τόνωση και την πρόθεση των επενδύσεων. Όχι όμως να λέμε ότι αυτό είναι τροχοπέδι και εμπόδιο για την πραγματική ε, υλοποίηση επενδύσεων στις επιμέρους χώρες. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γκαμπριέλε Μπίσοφ, ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε... Παρελθόν υπήρξαν ανισορροπίες μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν η οικονομική διακυβέρνηση τώρα να ευθυγραμμιστεί με τους κοινωνικούς στόχους της συνθήκης. Όπως είπε και η εκλεγήσα πρόεδρος Ursula von der ήρθε η ώρα να συμφιλιώσουμε ε, το κοινωνικό και το οικονομικό σκέλος της αγοράς. Πώς λοιπόν θα ενισχύσετε την κοινωνική διάσταση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τι προτίθεστε να κάνετε για να έχουμε μια καλύτερη σύγκληση προς τα πάνω, γιατί αυτό είναι ο απότερος στόχος. Θα προτείνετε νομοθετικές διατάξεις για να έχουμε αιτήσια αξιολόγηση των, ε, ε των, της πορείας των μισθών, της κάλυψης από συλλογικές συμφωνίες, ε, του εισοδηματικού κενού, και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπίσοφ, εγώ και με βάση την προσωπική μου πείρα, γιατί διατέλεσα και πρωθυπουργό. Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε καταρχήν συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για τις οικονομικές μας επιλογές και μαζί με τον συνάδελφο Νίκολα Σμιτ αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Να συνεργαστώ με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες μας. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου άρχισε την τελευταία διετία να περιλαμβάνει πολύ σοβαρά και την κοινωνική διάσταση. Και αυτό ήταν κυρίως απόρρια της απόφασης του Γκέτεμπορκ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Και σήμερα θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση και πέραν της συμφωνίας του Γκέτεμπορκ. Και αυτή ήταν και η εντολή που έλαβα στην ανάθεση καθηκόντων μου. Να συμπεριλάβω δηλαδή και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως ξέρουμε όλοι, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν μία ισχυρή κοινωνική διάσταση και όχι μόνο μία ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση. Και αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι το νέο εργαλείο για να δώσουμε στα κοινωνικά ζητήματα την προτεραιότητα που αξίζουν. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλληλο νομικό εργαλείο, το κατάλληλο νομικό μέσο για να, συνδέσουμε και την, να το συνδέσουμε με την πρωτοβουλία για το κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Χαίρομαι πάντως που τονίσατε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Συγκεκριμένα όμως, τι θα κάνετε για να ενισχύσετε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά και συμφωνώ με την πρόταση για τον κατώτατο μισθό δεν την ανέφερα γιατί δεν εμπίπτει άμεσα στο χαρτοφυλάκιό μου, αλλά στο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα στηρίξω την πρόταση για τον κατώτατο μισθό. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, θα πρέπει να εμ, κινητοποιήσουμε και το κοινό, να δημιουργήσουμε μια ευαισθητοποίηση ώστε και στα κράτη-μέλη να εμπλέξουμε τους κοινωνικούς εταίρους και στον εθνικό δημόσιο διάλογο. Ή ανάμειξη των κοινωνικών εταίρων θα εμπλουτίσει το διάλογο και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικοινωνήσει καλύτερα με τα κράτη-μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους ε, τις αποφάσεις της κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο κύριος Λούντε Κνίτερμαϊερ από το ΕΛΚ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνι. Πίσω σας κάθομαι, βλέπω ε, κοιτώ πάνω από τον νόμο σας. Αυτό κάνει το Κοινοβούλιο κατά καιρού. Ε, σα ελέγχει δηλαδή. Ε, αφιερώσατε το μεγαλύτερο μέρος των γραπτών απαντήσεών σας ε, στην φορολογία. Αναφερθήκατε στην ψηφιακή φορολογία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με ε, δύο άλλες προτάσεις ε, που έχει δει με ευνοϊκό μάτι στο παρελθόν το Κοινοβούλιο. Η μία είναι για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιριών και η άλλη είναι για το ΦΠΑ. Τι συγκεκριμένα βήματα θα αναλάβετε για να ξεμπλοκάρουν αυτές τις προτάσεις στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάγερ. Δεν ξέρω να κοιτάω εσάς ή τους, ή τους άλλους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και η κοινή ενωπημένη φορολογική βάση των εταιριών είναι δύο βασικά ζητήματα ε, που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο για τη φορολογία. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για, ε, ε, του ΦΠΑ, Νομίζω ότι πρόσφατα είχαμε σχετικές αποφάσεις ιδιαίτερα. Την πρόταση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce. Και η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα είναι πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη στο εγγύς μέλλον. Η γενική πρόταση για αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο θα προωθήσω, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις που αποφασίσαμε πρόσφατα απαιτούν άμεσα την δέσμευση των κρατών μελών. Δεν είναι λοιπόν η άμεση προτεραιότητά μου το ΦΠΑ, ίσως μετά από κάποια τρίμηνα, εντό του 2020 να ασχοληθώ. Όσον αφορά την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιριών, αυτή είναι απόλυτη προτεραιότητα, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Είναι κάτι που συνδέεται και με τις συζητήσεις στο πλαίσιο του ΩΣΑ. Εγώ προσωπικά πάντως δεν θα περιμένω και θα προτείνω να προχωρήσουμε πάνω στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μου. Η επερώτησή μου έχει να κάνει με τον συνοριακό φόρο άνθρακα, διότι είναι πολύ σημαντικός για το δίκαιο εμπόριο. Πόσο καιρό Νομίζετε ότι θα χρειαστεί η πρόταση αυτή, λαμβανομένου υπόψη ότι από τεχνική φύση είναι δύσκολη. Και πότε νομίζετε ότι ε, θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Ε, όσον αφορά τον συνοριακό φόρο άνθρακα. Όλοι γνωρίζουμε τους ε, τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε. Αυτό όμως ε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το μέτρο προσαρμογής ε, μπορεί να είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Χωσέ Γκούσμαου από την Γκούε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ είμαι πίσω σας, ορίστε, Επίτροπε. θα ήθελα να συζητήσουμε το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο ενεργή στο να πιέζει τι οικονομίε που είχαν προβλήματα χρέου και ελλείμματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά αυτέ που είχαν πλεονάσματα και περιθώριο δημοσιονομικό η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μεγάλη πυγμή και ήταν πολύ ταχεία στο να ζητήσει πίσω επιστροφές από το να ζητήσει επενδύσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται να υπήρξε επιβράδυνση, μάλλον υπερβολική επιβολή αυστηρότητας στις οικονομίες με προβλήματα. Όμως με μακροοικονομικές ανισορροπίες συστηματικά στην ε, νομισματική και οικονομική μας πολιτική δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι μακροπρόθεσμα. Πρέπει να δούμε το σκέλος των επενδύσεων στον υπολογισμό του ελλείμματος. Θα ήθελα εδώ να ξέρω την άποψή σας και τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τα συστηματικά συστηματικά τα διευθυντικά πλεονάσματα που έχουν παρατηρηθεί ε, και αυτό βάσει των γραφειοκρατικών. Των, ε, της αιτήσεως για την ανάπτυξη. Ε, κύριε Κουσμάου, έχουμε τους κανόνες μας. Οι κανόνες μας αλλάζουν ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον και το τι συμβαίνει στην ε, παγκόσμια οικονομία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η οικονομική μας πολιτική είναι πάντοτε απαράλλαχτη. Ε, οπωσδήποτε η κρίση που γνωρίσαμε ήταν βαθιά πριν από 10 χρόνια. Και μάλιστα διαρκείας. Η βαθιά αυτή, αυτή κρίση προκάλεσε τεράστια προβλήματα χρέους σε πολλές χώρες και αυτό είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες, της τις μέρημνες της οικονομικής μας πολιτικής. Πιστεύω ότι ήμασταν σχετικώς αποτελεσματικοί στο να χειριστούμε τα ελλείμματα και να διατηρήσουμε σε σταθερό επίπεδο το χρέος. Α, όχι όμως να το μειώσουμε και δραστικά. Τώρα αντιμετωπίζουμε και όλο ένα κατανοούμε καλύτερα το βαθμό του προβλήματος. Έχουμε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, διότι ο ρυθμός επιβραδύνεται και δεν ξέρουμε σε τι βαθμό και για πόσο. Υπ' αυτήν την έννοια, οι οικονομικές μας πολιτικές θα πρέπει να έχουν ένα σαφή προσανατολισμό για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις και να ζητήσουμε σε όσους έχουν ε, περιθώριο στον προπολογισμό τους να το αξιοποιήσουν για να ξαναρχίσει η ανάπτυξη. Δεν λέμε να αλλάξουμε τους κανόνες, λέμε να τους προσαρμόσουμε στις μεταβολές ε, του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επερώτηση. Ναι, αλλά ένα από το πρόβλημα των οικονομιών που είναι υπερχρεωμένε είναι ότι κάθε χρόνο ένα μέρο ε, του δημοσιονομικού ωφέλου ε, του εισοδήματο θα πρέπει να υποβληθεί για επιστροφέ σε άλλε οικονομίε εντό εντός, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων φορέων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλων ε, οικονομιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τον ανταγωνισμό. Όμω, θα πρέπει με του χαμηλού συντελεστέ, τα χαμηλά επιτόκια που πρόβλεψε η ΕΚ, να πούμε ότι προσπάθησε να λύσει ένα μέρο του προβλήματο. Εσεί θεωρείτε ότι η πραγματικότητα αυτή είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε στα πλαίσια του 116 ή μάλλον με το 116 να χρησιμοποιήσετε τους κανόνες της ΕΚΤ για τα χαμηλότερα επιτόκια στην περίπτωση του και να δημιουργήσετε μια κοινή φορολογική εταιρική βάση που να μην είναι σε χαμηλά επίπεδα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει χαμηλών ε, διαφορετικών μάλλον φορολογήσεων στις εταιρείε. Θα προχωρήσουμε με την πρόταση αυτή, χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εργαλεία που διαθέτουμε. Με τις δυσκολίες που τις γνωρίζουμε βέβαια, αλλά και με πολιτική ε, ε, αποφασιστικότητα, με πολιτική πυγμή Κοινοβούλια και Επιτροπή μαζί. Σας ευχαριστώ. Ο Ρόμπερτ Μπιέντρον έχει το λόγο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Είναι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν ο επόμενος. Έχω τον κύριο Μπιέντρον στον κατάλογο. Καλώ. Ντέμιον Μπουσελάγκερ από την Επιτροπή Προπολογισμών, μέλο των Πρασίνων. Ο συνάδελφο έχει λάβει τη θέση του κύριου Μπέντρον. Τζον Χάουαρθ από το Ηνωμένο Βασίλειο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και το ανέφερε και ο κατάλογος. Okay, ε, ε, Καλώς, ζητώ συγγνώμη. Δεν το γνωρίζαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, στην επιστολή ανάθεση καθηκόντων η εκλεγής επιτροπός σας ανέθεσε την θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου για το, και το συντονισμό του μελλοντικού προγράμματος InvestEU. Ταυτόχρονα, ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης θα αναλάβει το συντονισμό του έργου του επενδυτικού σχεδίου για τη βιώσιμη Ευρώπη με στόχο της, την προσέλκυση επενδύσεων ενός τρισεκατομμυρίου για το περιβάλλον στην επόμενη δεκαετία. Ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θετία το Συμβούλιο είχε καταλήξει μερική συμφωνία για το InvestEU. Πώς ε, θα διαχωρίσετε τις ευθύνες σας με τον κύριο Ντομπρόφσκι σε ό,τι αφορά το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και ποια θα είναι τα αποτελέσματα και συνέπειες του νέου ε, επενδυτικού σχεδίου ε, των βιώσιμων επενδύσεων στο πρόγραμμα InvestEU. Σας ευχαριστώ κύριε Χόρθ. Γενικώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να συντονιστούμε, να συντονίσουμε το έργο μας. Και έχουμε διαφορετικά εργαλεία και μηχανισμούς. Έχουμε καταρχήν το πρόγραμμα InvestEU. Το InvestEU το έχετε ήδη συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το InvestEU έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Θα έχουμε τώρα και μια ισχυρή τεχνική ικανότητα σε αυτό το κόμπο που δημιουργεί το InvestEU. Αλλά θα είναι πολύ χρήσιμο να προωθήσουμε και τις επενδύσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Ευρώπης. Οπότε θα συμπορευτούμε με τον κύριο Ντομπρόφσκης. Θα συνεργαστούμε, αν και εκείνος είναι πιο ειδικό στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στα πλαίσια του σχεδίου ε, για τις ε, βιώσιμες επενδύσεις στην Ευρώπη. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στον προσδιορισμό του σχεδίου και την πρόθεση του προγράμματος InvestEU. Χρειαζόμαστε πολλούς μηχανισμούς και μέσα για να μοχλεύσουμε επενδύσεις. Θα χρειαστούμε πολλές επενδύσεις και για τη βιώσιμη Ευρώπη και για την οικολογική μετάβαση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, επερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, απλή επερώτηση. Εγώ θα ελπίζα όλες οι επενδύσεις που γίνονται στα κοινοτικά προγράμματα να είναι φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις και βιώσιμες επενδύσεις. Εσείς, ποιο πιστεύετε θα είναι ο βασικός μηχανισμός για να εξασφαλίσουμε φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις και στα πλαίσια του προγράμματος InvestEU, αλλά και στα υπόλοιπα προγράμματα. Τζεντιλόνι. Ναι, έχουμε μια μεθοδολογία για να θωρακίσουμε περιβαλλοντικά τα μέτρα μας. Είναι κάτι σχετικά πρόσφατο στις υπηρεσίες μας. Εξετάζουμε πάντα την περιβαλλοντική διάσταση όλων των επενδύσεων. Στο InvestEU, για παράδειγμα, έχουμε τις επενδύσεις στις υποδομές που στόχο έχει την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και όλες οι λοιπές πτυχές των επενδύσεων και για τις προτεραιότητες του InvestEU είναι ε, περιβαλλοντικές, ε, ε, ψηφιακές, κοινωνικές διατάξεις, ε, παιδεία, ε, δεξιότητες, βιώσιμες υποδομές και σίγουρα η περιβαλλοντική διάσταση θα συνοδεύεται από μια σαφή μεθοδολογία. Ντάμιεν Μπέσελάγκε συγγνώμη, από την Επιτροπή Προπολογισμών και του Πράσινου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Οι νέοι επλήγησαν ε, πολύ σκληρά από την τελευταία οικονομική κρίση. Πολλοί δεν κατάφεραν να βρουν την πρώτη τους δουλειά, το οποίο είχε και σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ε, σχετικά με το πρώτο πιθανό όργανο του προϋπολογισμού μας ε, για την σύγκληση. Ε, όσον αφορά το μέγεθος και την ευελιξία του εργαλείου αυτού. Θα επιτρέψετε να πάνε τα χρήματα εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο και δεύτερον θα επιτρέψετε την ε, χρήση ε, μηχανισμών ώστε να αυξηθεί η ε, ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης και τρίτον σχετικά με την μακροοικονομική σταθεροποίηση ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, νομίζω ότι... Η πρόταση που ε, που επιβεβαιώθηκε, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο στην διάσκεψη κορυφής σχετικά με αυτό το νέο εργαλείο για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το BICC για τη σύγκληση νομίζω ότι είναι χρήσιμο και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς και να θεωρηθεί και εργαλείο σταθεροποίησης. Γνωρίζουμε ότι η συζήτηση για ένα τέτοιο εργαλείο πάντα ήταν δύσκολη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω όμως ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ στοχευμένη και στόχος είναι να ενισχυθούν ε, διαθροτικές ε, μεταρρυθμίσεις και η σύγκληση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει σοβαρή χρηματοδότηση καθώς και παρακολούθηση στη συνέχεια. Αυτή είναι προσωπική μου δέσμευση απέναντι στην Επιτροπή σας. Επερώτηση. Πώ βλέπετε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Προϋπολογισμού όσον αφορά την διακυβέρνηση, ε, την απαλλαγή του BICC και θα συμπεριλάβετε και ε, κριτήρια για το κλίμα. Ναι, θα συζητήσουμε μαζί τα κριτήρια διακυβέρνησης και τις προτεραιότητες αυτού του εργαλείου. Σίγουρα θα λάβουμε υπόψη σοβαρά το κλίμα ως προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Δράγος από um, There Φαίνεται ότι υπάρχει γενική συνένεση ότι οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι κρίσιμε και έχουν μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την αθεκτικότητα στου κραδασμού. Βέβαια, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει επιβραδύνει τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που χαρακτηρίστηκε από ένα αίτημα σταθερότητας και μια κόποση των μεταρρυθμίσεων. Αυτά θα πρέπει να αλλάξουν όμως, ε, ε, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή δικά δηλαδή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ε, χώρες εκτός του ευρώ χρήζει προσοχή. γιατί υπάρχουν μεγάλες δεσυνδέσεις μεταξύ των, οικονομικών, των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλληλένδετες οι οικονομίες, οπότε οι, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εκτός της ευρωζώνης δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την ανταγωνιστικότητα και πιο μακροπρόθεσμα, ενώ το κοινωνικο-οικονομικό κόστος θεωρεί, ε, κρίνεται συνήθως βράχη πρόθεσμα. Για τις δεξιότητες, για τη μεταρρύθμιση ε, στην παιδεία, στην υγεία ή στην εξάλληψη της φτώχειας, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από ένα πρόθεσμο κόστος. Ε, συμφωνείτε με αυτή την προοπτική και ο εσείς ως πρωταθλητής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα στηρίξετε προστάσεις τις προθέσεις ε, των ε, χωρών μελών εκτός της Ευρωζώνης να εφαρμόσουν ε, με γοργό ρυθμό τα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τους. Ευχαριστώ κύριε Πισλάρου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστερνιζόμαστε το στόχο της πρόθεσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την προτεραιότητα. Γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια οικονομική επιβράδυνση με πολλούς τρόπους. Μπορεί να έχουμε πιο ανοιχτές ή χαλαρές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι μεσοπρόθεσμα ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μας, λοιπόν, και σε όλες τις ε, νομοθετικές μας διατάξεις, αν χρειαστεί να αλλάξουν, θα δοθεί προτεραιότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και γνωρίζετε κι εσείς που είστε αιρετοί, ότι πολύ συχνά αυτή η κόποση απέναντι στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν οφείλεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά σε κάποια εθνικά στοιχεία, σε κάποιους εθνικούς παράγοντες ή εθνικούς λόγους. Αστάθεια, για παράδειγμα. Η αστάθεια, ακριβώς για, το, για τους λόγους που αναφέρατε, λαμβάνεται υπόψη. Γιατί αποφασίζουμε κάτι που δεν θα έχει συνέπειες βραχυπρόθεσμες, αλλά μακροπρόθεσμες, οπότε η πολιτική αστάθεια ενισχύεται στις χώρες μας. Και αυτή η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει την τάση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ή την ενασχόληση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτός όμως είναι ένας λόγος παραπάνω για τα θεσμικά όργανα να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να δείξουν μεγαλύτερη προσήλωση σε αυτό το στόχο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Επερώτηση έχετε? Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα InvestEU επανειλημμένως και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε θα πρέπει να έχουμε πιο απλή, αποτελεσματική και εύχριστη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού παρά τους περιορισμούς. Το θέμα της τεχνικής αρρωγής θα το χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τις γεωγραφικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατομελών και να έχουμε η ισότιμη, ακριβωδή και η γεωγραφική κατανομή των ε, διαφόρων κονδυλίων δεδομένων των διαφορετικών χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα ότι ένα τόσο σημαντικό σχέδιο για μας, όπως είναι το πρόγραμμα InvestEU, που στόχο έχει να γύρει περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αδιανόητο να περιορίζεται σε μερικές μόνο περιφέρειες ή σε μερικές μόνο χώρες. Οπότε, η δέσμευσή μου είναι να έχουμε μία ακριβοδίκαιη κατανομή, ισότιμη κατανομή ε, του σχεδίου Invest EU σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε ο κύριος Διόρη από το ΕΛΚ. Η κυρία Διόρη. Ε, με... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αν επιτρέπετε θα μιλήσω ουγγρικά. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Ξεκινήσατε λέγοντας ότι είναι καθοριστική η εμπιστοσύνη. Μπορείτε να μας πείτε αν στα πλαίσια του ρόλου σας θα είσαστε πραγματικά αξιόπιστος και αν θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της Ιταλίας. Ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει κυρώσεις οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και μάλιστα στα διαρθρωτικά ταμεία η Ιταλία πήρε και έκπτωση. Ε, εγώ εκπροσωπώ την Ουγγαρία, μια χώρα η οποία απειλήθηκε με αναστολή των πληρωμών από τα, από τα Ταμεία Συνοχής. Και στην χώρα μου επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά λοιπόν το δύο, σύστημα αυτό των δύο μέτρων και δύο σταθμών στην χώρα εφαρμόστηκαν διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα πολύ γρήγορα. Εσείς ως Επίτροπος, τι θα κάνετε για το σύστημα αυτό των δύο μέτρων και δύο σταθμών, πώς θα το αντιμετωπίσετε και τι θα κάνετε και ε, προς όφελος των χωρών που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκιόρη. Είναι απόλυτα σαφές για μένα ότι δεν θα έχουμε δύο μέτρα και σταθμά στην εφαρμογή των κανόνων μας. Είναι θέμα εμπιστοσύνη, καταλαβαίνω. Από αυτά που είπα το πρωί μπορείτε να το καταλάβετε, μπορείτε να δείτε και το βιογραφικό μου, αλλά πέραν αυτού είναι και θέμα εμπιστοσύνη. Είναι δέσμευση που αναλαμβάνω. Δεν θα υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Και είναι και προσωπικό μου ε, πεπραγμένο θα έλεγα από την θητεία μου στην Ιταλική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Πάντοτε προασπιζόμουν ακόμα και σε καιρούς όπου δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα στη χώρα μου, πάντοτε υπερασπιζόμουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ακόμη και αν έπρεπε να ασκήσω πίεση και στα πλαίσια αυτών των κανόνων να υπάρχει μια στάση που να ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη. Αυτό ήταν ανέκαθεν η θέση μου. Mm. Όχι δίπλα μέτρα και σταθμά ε, εις βάρος ιασδήποτε χώρας και εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να εργαστούμε για ένα κοινό σκοπό για το ευρώ. Επερώτηση. όμως η δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πλήττονται κυρίως οι επενδύσεις. Αλλά αν δεν υπάρξουν επενδύσεις θα έχουμε και αντίθετε συνέπειες. Και όμως σε κάποιες χώρες παρά την ε, ε, δυνατότητα παρά τις δυσκολίες τους, κατάφεραν να κάνουν καλά τα μαθήματά τους και να ξεφύγουν από το πρόβλημα της ενεργείας. Ενώ σε άλλους, ενώ η ενεργεία ήταν πιο χαμηλή, χρειάστηκε εξωτερική παρέμβαση. Εδώ λοιπόν πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας προσφέροντας ευνοϊκότερες συνθήκες στις επιχειρήσεις μας. Αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση υγείας των ευρωπαϊκών εταιριών και πώς θα προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε λοιπόν για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παρά τα μετά που προβλέπονται. Ναι, έχουμε πολλά εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό. Ένα για παράδειγμα θα είναι το Συμβούλιο ε, για το φόρο στον άνθρακα για να αποφύγουμε τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για εις βάρος εταιριών. Το άλλο θα είναι ο ενιαίος εταιρικός φόρος και πολλά πολλά άλλα. Δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος για... και αρνητικός για το ότι πετύχαμε. Σε σχέση με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανεργία τα τελευταία χρόνια. Διότι το πρόβλημα σαφώς υφίσταται σε πολλές χώρες, ιδίως τη δική μου και συγκεκριμένα σε ειδικέ περιοχές. Εάν όμως δείτε τι γινόταν στα χρόνια της κρίσης, έχουμε προοδεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο ως εφαλτήριο και να πάμε σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους ε, και τον ε, υποψήφιο επίτροπο κύριο Τζεντιλόνι για τις απαντήσεις του. Τώρα θα καλέσω τον κύριο Τζεντιλόνι να κάνει μια σύντομη πεντάλεπτη καταληκτήρια παρέμβαση πριν ολοκληρώσουμε και την ακρόαση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ. Είχαμε τρεις ώρες για να συζητήσουμε, να συζητήσουμε εντατικά. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που όπως ε, έμαθα τα τελευταία χρόνια είναι υψηλού επίπεδου και μου επέτρεψε να εργαστώ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο θεωρούμε ότι σήμερα περάσαμε σε μια πολύ σημαντική, ε, από μια πολύ σημαντική φάση της δημοκρατικής διαδικασίας. Συχνά γίνεται λόγος για την ε, ικανότητα του δημοκρατικού συστήματος, για το πόσο είναι πλήρες και εδώ Σας διαβεβαιώ ότι για να προετοιμαστώ για την ακρόαση αυτή και να είμαι σε θέση να πάρω μέρος απαντώντας τις ερωτήσεις σας, ήταν ακριβώς ε, η επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού. Η δημοκρατία στην Ευρώπη μπορεί να έχει και κάποια όρια, αλλά και υπαρκτή είναι και λειτουργεί και είναι ένα asset, ένα στοιχείο του ενεργητικού, στο οποίο πρέπει να ποντάρουμε για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος στο μέλλον στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά. Ε, ένα σημείο θέλω να τονίσω όλος ιδιαίτερος. Σε ένα σημείο θέλω να είμαι σαφέστερο, σαφέστερος, γιατί με την πάροδο των ερωτήσεων κάποια πράγματα επαναλήφθησαν ε, συχνά και κάποιες ερωτήσεις προσωμίαζαν μεταξύ του. Το βασικό σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ λοιπόν είναι ότι θα προσπαθήσω να μην άθεθω σε καταστάσεις ε, τέλματος, σε καταστάσεις μη προόδου. Για να το πετύχω αυτό θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το επιτρέπουν οι κανόνες μας, την συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μπούμε σε κατάσταση τέλματος δεν μπορούμε να μην πάρουμε αποφάσεις για πολλά από τα θέματα που μας απασχόλησαν από το πρωί. Τους φόρους, την ε, τοποθέτησή μας απέναντι στο θέμα ανάπτυξη, τους κανόνες που διέπουν τους προπολογισμού και τόσα άλλα θέματα που είναι και ενδεχομένως εκτός του χαρτοφυλακίου μου δεν πρέπει λοιπόν να αφαιθούμε σε τέλμα και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε ένα μόνο εργαλείο. Με δύο λόγια το λέω. Πολιτική και εμπιστοσύνη. Χωρίς πολιτική, χωρίς να προσπαθήσουμε να δημιουργούμε συμμαχίες, να συμφωνούμε μεταξύ διαφορετικών ομάδων, να μην αποδεχόμαστε τον διαχωρισμό βοράς εναντί νότου, Ανατολή απέναντι στη Δύση και άλλων περιοχών της Ευρώπης. Χωρίς λοιπόν την πολιτική διάσταση δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το τέλμα. Και επίσης χρειαζόμαστε και εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν θα υπάρχουν ε, νικητές και ιτημένοι. Ε, Μόνο η ήττα του κοινού μας ε, ευρωπαϊκού εγχειρήματο θα υπάρξει χωρίς εμπιστοσύνη. Γι' αυτό σας ζητώ εμπιστοσύνη. Είμαι Ιταλός. Ανήκω στην οικογένεια των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Εάν όμως επιβεβαιωθώ ως Επίτροπος για τις οικονομικές υποθέσεις, θα είμαι ένας Επίτροπος της Οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Ε, Πραγματικά θα είναι η πατρίδα μου και το πεδίο δράση μου η Ευρώπη. Γι' αυτό σας ζητώ εμπιστοσύνη. Ζητώ την στήριξή σας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε αρμονικότατα στο... για τα κοινά μας ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ για το σημερινό πρωινό και σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Τζαντιλόνη. Και τώρα κυρίσω τη λήξη της ακρόασης. Συνεδρία των συντονιστών θα γίνει και κλεισμένο των θυρών για την αξιολόγηση της ακρόασης. Ευχαριστώ.